έστειλα ένα υπόμνημα ε, μίας ε, οργάνωσης υπέρ των καταναλωτών και υπάρχει ε, η εγκατάλειψη της θύρας της, γκρίζια, της γκρίζας φώκες διότι δεν υπάρχει τέτοια ζήτηση. Άρα και η απαγόρευση μπορεί να έχει επιπτώσεις. Τέλος, αναφέρθηκε από το ΕΛΚ από τον Ανδρέας ότι θα πρέπει να είμαστε συμβατοί με τις προδιαγραφές του ΠΟΕ και η συμφωνία του ΓΚΑΤ επιτρέπει στα κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη του ΓΚΑΤ να λάβουν αποφάσεις με βάση την ιδιάζουσα κατάστασή τους. Άρα είναι αδιέξοδο το θέμα της σήμανσης. Θα πρέπει να έχουμε την ε, μεγαλύτερη δυνατή απαγόρευση εξαιρώντας την θύρα των Ινουίτ. Πρόεδρος, η Επιτροπή ίσως θα ήθελε να λάβει το λόγο σε αυτή τη φάση, αλλά επειδή δεν ήμουν εδώ στην ακρόαση, κοίταξα μόνο τα υπομνήματα και τις παρουσιάσεις της εισηγής. Νομίζω ότι ο κύριος Μάρτιν αναφέρθηκε σε κάτι που θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ πρέπει να σας υπενθυμίσω τι μας ζητείτε εδώ για την εσωτερική αγορά, διότι δώσαμε συνεχή μάχη με την Επιτροπή Γεωργίας, γιατί θεωρήσαμε ότι δεν είναι θέμα που αφορά την ευημερία των ζώων. Άρα ο κύριος Μάρτιν έχει δίκιο. Παράλληλα με αυτά που κάναμε για την ε, οδηγία που αφορά τα, την, το τρίχωμα της γάτας και του σκύλου το οποίο τίθεται σε εμπορία, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαγόρευση στην ε, ε, εσωτερική αγορά καθώς και η διαμετακόμιση και οι εισαγωγές. Εκεί λοιπόν που γίνεται η θύρα της φώκιας που αφορά αυτόχθονες πληθυσμούς σε ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να δούμε πώς θα επιτρέψουμε σε αυτό να συνεχιστεί με βάση την ε, ευζοία αυτού του είδους αλλά βεβαίως ε, δεν μιλάμε για εμπόριο το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να το έχετε αυτό υπόψη, αλλά εγώ δεν θα αποφασίσω αυτό που θα αποφασίσετε εσείς. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Έχουν ακουστεί διαφορετικές απόψεις Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ, κατά, τι θα γίνει με την επισήμιση, με την πλήρη απαγόρευση, είναι συμβατή με τις ε, προδιαγραφές του ΠΟΗ και ούτω καθεξής. κυρία θα παρέμβετε στο τέλος. Θα μας μιλήσει η Επιτροπή καταρχή, ο κύριος Λάγκεντορφ. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω λίγα γενικά σχόλια για τα όσα συζητήθηκαν μέχρι τώρα. Το θεμελιώδες ερώτημα που καθοδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τούτη εδώ τη συζήτηση τον τελευταίο 1,5 χρόνο όταν δηλαδή συντάσαμε την πρόταση ήταν τι πρόκειται να λειτουργήσει τι μπορεί να λειτουργήσει με ορισμένους αντικειμενικούς σκοπούς που επιθυμούμε να επιτύχουμε, ε, κυρίως θέματα προστασίας των ζώων βέβαια. Το συμπέρασμά μας μετά από την διεξαγωγή ορισμένων μελετών και έχοντας ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι εν τέλει ότι ούτε η πλήρης απαγόρευση, ούτε ένα σύστημα επισήμανσης που να ακολουθεί περίπου αυτά που λέει η κυρία Γόλη στο σχέδιό της δεν θα λειτουργήσουν, δεν θα αποδώσουν. Πλήρης απαγόρευση δεν θα επιτύχει διότι δεν θα έχει επαρκή βαρύτητα στις ε, χώρες μέλες ούτε και στις υποψήφιες χώρες μέλη ώστε να τις αναγκάσει να ε, βελτιώσουν τα μέτρα προστασίας των ζώων. Θεωρούμε και γι' αυτό εξετάσαμε την επιλογή αυτή στο Impact Assessment ότι ένα σύστημα επισήμανσης όπως περίπου το προτείνει η η ούτε και αυτό πρόκειται να αποδώσει, να επιτύχει τον σκοπό. Πιστεύουμε ότι για τον λόγο εάν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα θα έχουμε ποικιλία σημάτων τα οποία ε, θα ε, επιτίθενται στα προϊόντα από την θύρευση της φώκιας, τα οποία θα οδηγήσουν σε σύγχυση ε, τους καταναλωτές και δεν θα επιτρέψει έτσι να ασκηθεί πίεση στις χώρες ώστε να αλλάξουν τις πρακτικές που ακολουθούν. Σχετικά με τις εξαιρέσεις υπέρ των Ινουίτ. Αυτοί εξαιρούνται βέβαια από την απαγόρευση ώστε δεν χρειάζεται να ζητήσουν ειδική εξαίρεση όπως άλλωστε και εσείς είχατε ζητήσει στην δήλωσή σας, αλλά και σύμφωνα με τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο πρόεδρος Μπαρόσο απέναντι σε εκπροσώπους των κοινοτήτων Ινουίτ. Δεν θεωρούμε ότι θα ήταν είτε σωστό είτε επιθυμητό να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης των Ινουίτ με κάποιο τρόπο και ιδίως ο λόγο των κοινωνικο-οικονομικών συμφερόντων που προστατεύουμε αυτή τη στιγμή με τον τρόπο αυτό. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να, εξαιρε... να ε, περιοριστεί η εξαίρεση υπέρ των Ινουίτ, μειώνοντας για παράδειγμα την δυνατότητα εμπορίας ορισμένων προϊόντων φώκιας. Θεωρούμε ότι είναι σωστή η ιδέα να εξεταστούν οι ορισμοί, εξετάζοντας και τι λέει το ICC. Είμαστε υπέρ λοιπόν της εξέτασης αυτής, αλλά μόνο εάν προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τις έννοιες, όχι όμως να περιορίσουμε τις εξαιρέσεις. Αυτή είναι η θέση μας. Μια τελική παρατήρηση για, το, ε, για την θύρευση μικρής κλίμακας που δεν νομίζουμε ότι μπορεί να εξαιρεθεί από την πρόταση και ε, οι λόγοι έχουν αναφερθεί σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα προβλήματα που θα τεθούν ε, υπό την ισχύ των διατάξεων του ΠΟΕ για μη ε, διακρίσεις κλπ. Υπάρχει και μια ε, διάταξη που προβλέπει ιδιαίτερες συνθήκες σε ορισμένες χώρες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άρα υπάρχει μια διάταξη η οποία θα επέτρεπε στην διαδικασία εξέτασης αιτήσεων εξαιρέσεως να εξεταστούν οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες οι οποίες θα περιλαμβάνουν και την θύρα μικράς κλίμακας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να αποκριστεί ούτε και καλή ιδέα είναι μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ και θα αφήσει επικίνδυνα παράθυρα στην νομοθεσία. Διότι κάτι που μπορεί να είναι μικρά κλίμακα σήμερα μπορεί να γίνει κατάχρησή του αύριο. Θα ήμασταν λοιπόν κατά της εξαίρεσης της ε, θύρας μικράς κλίμακα από τις προτάσεις και νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε πολύ περισσότερο με την κυρία Ουάλης δηλαδή να ληφθεί υπόψη η ε, θύρα μικράς κλίμακας και όχι να εξαιρεθεί όπως έχουν, να αποκλειστεί όπως έχουν ε, ε, ζητήσει ορισμένοι. Και το θέμα της νομικής βάσης επίσης 95 στο επεξηγηματικό μνημόνιο επανερχόμαστε στο ερώτημα αυτό που τέθηκε και στη διάρκεια της ακρόασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταλληλότητα του άρθρου 95 ως νομικής ε, βάσεως έχει εξηγηθεί η θέση μας στο υπόμνημα και εν μέρη ε, τουλάχιστον απαντούμε στις ερωτήσεις σας εκεί. Δεν θυμούμε ακριβώς σε ποια σελίδα, θα βρείτε όμως τις εξηγήσει και αναφερόμαστε και σε ε, αποφάσεις του δικαστηρίου. Νομίζω ότι όλοι κάνατε σαφείς παρεμβάσεις. Η πρόκληση τώρα για την κυρία Γουάλης είναι να αναζητήσει και να επιτύχει κάποιο συμβασμό. Εσείς τώρα. Επανέρχομαι πρόεδρε. Προσπάθησα να συντάξω μια έκθεση η οποία ήταν επίγουσα και προσπάθησα να θέσω ορισμένα επιχειρήματα και να εκφράσω ορισμένες ανησυχίες αναφέρομαι και στην ενιαία αγορά και μάλιστα εκτεταμένα. Είσαι οι ανησυχίε μου ότι όντως αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο κατακαιρματισμού γιατί διάφορες χωρίς μέλη κάνουν διαφορετικά πράγματα. Προσεγγίζοντα όμως ε, το αντικείμενο με, ε, με απαγόρευση γιατί είναι διαφορετικό από ότι για τις γούνες σκύλων και ε, γάτων. δεν είναι η ίδια περίπτωση όπως με, τις, ε, με, το δέρμα Δεν υπάρχουν δηλαδή ε, προϊόντα τα οποία θα υποφεληθούν από την απαγόρευση και επομένως θα στρεβλώσουν την αγορά. Θυμίζω και τα σχετικά με την διαφήμιση του καπνού. Αναφέρομαι λοιπόν σε θέματα ενιαίας αγοράς και θέτω θέματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν και που θα πρέπει να τα έχουμε στη σκέψη μας ως Επιτροπή. Κατανοώ τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ίδια πράγματα ε, σκέφτομαι και εγώ, όπως και αυτή η Επιτροπή δηλαδή, επί πολύ περισσότερο χρόνο. Λένε ότι οι ετικέτες, η επισήμανση μπορεί να οδηγούν σε σύγχυση. Μας δόθηκε ένας μήνας για να συντάξουμε ένα σχέδιο για ε, ένα σύστημα επισήμανσης, τουλάχιστον αναγνωρίστε ότι κάναμε μια προσπάθεια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα εάν κληθώ να, εργαστώ με, να συνεργαστώ με συναδέλφους που θα βασίζουν τις ιδέες τους ε, στην δήλωση για την βελτίωση των δικαιωμάτων των ζώων, προστασία των ζώων κλπ. καθώς και προστασία ορισμένων ηθαγενών πληθυσμών. Ευχαρίστω το πράξω, αλλά είναι σαφές από τα όσα συζητήσαμε σήμερα ότι υπάρχει και ένα μέρος που, ε, των συναδέλφων θα ήταν υπέρ ενός συστήματος ε, επισημάνσεως. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν προς τα που κινούνται οι τάσεις, αλλά βεβαίως είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ με άλλους συναδέλφους και βεβαίως εν τέλει είμαι απλώς η συγγετριά σας και ο ρόλος μου είναι το κείμενο, τα κείμενα που θα συντάξω να απηχούν τις απόψεις σας. και να καταδείξω ορισμένες από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε τέτοιου είδους νομοθετήματα. Και βέβαια πρέπει να το κάνουμε με τρόπο συνεκτικό και ε, προσεκτικό. Όταν λέτε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα, δεν είμαι βεβαίω ότι αυτό είναι σωστό. Γιατί στην περίπτωση αυτή λειτουργεί καλύτερα η αγορά. Τουλάχιστον ε, αυτή είναι η νομική ερμηνεία που δίνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα προϊόν το οποίο θα επωφεληθεί από μια ενδεχόμενη απαγόρευση. Πρόεδρος, εγώ ενδιαφέρομαι περισσότερο από την πλευρά του καταναλωτού. Δηλαδή, ε, οι εναλλακτικές επιλογές για ε, δέρματα ε, σκυλιών και γατιών είναι μάλλον συνθετικά. Ναι, μιλάμε για προϊόντα, όχι μόνο γούνα. Εξακολουθούμε να μιλούμε για προϊόντα. Αν και βέβαια κυρίως σκεφτόμαστε την γούνα. Εσείς τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να σας πω ότι κατανόησα ότι όλα τα παραδοσιακά προϊόντα που προέρχονται από την φώκια είτε είναι το λίπος είτε το δέρμα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν από άλλα προϊόντα. Άρα δεν υπάρχει αποκλειστικότητα προϊόντων που προέρχονται από τη φώκια. Ούτε για τον Καναδά, ούτε για την Ευρώπη. Καταρχήν και δεύτερον, κανένας ε, δεν διέψευσε τους εμπειρογνώμονες ε, σύμφωνα με τους οποίους τους αυτό πληθυσμούς, τα αποθέματα φώκιας ε, μειώνονται και ιδιαίτερα αυτό αφορά τις νέες φώκες, άρα υπάρχει μεγάλος ε, κίνδυνος εξάλληψης αυτού του είδους από τον πλανήτη. Τρίτον, μία καναδική ρύθμιση που αφορά την ε, παράνομη θύρα θα πρέπει να μας απασχολήσει, ιδιαίτερα όσο αφορά την εκδορά του ζώου. Αυτή η απόφαση έχει τηρηθεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν όμως συγκεκριμένες κυρώσεις για την κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της θύρας και ως προς την πλήρη απαγόρευση γνωρίζω ότι υπάρχουν χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουν αυτή την απαγόρευση και μέσα στα πλαίσια του κατακαιρματισμού της αγοράς εάν υπάρχουν χώρες που θέλουν να αγοράσουν το δέρμα φώκιας δεν χρειάζεται να την θυρεύσουν σε τόσο ευρία κλίμακα. Άρα η δημόσια ακρόασή μας έδειξε πώς έχουν τα πράγματα έμπρακτα και οι 425 βουλευτές αποφάνθηκαν καθώς και η θέση αυτή της Επιτροπής. Η κυρία Ρόιτοβα, ξέρω ότι έγινε μία ανταλλαγή απόψεων, υπάρχουν ε, τροπολογίες, η κυρία Γόλης θα προσπαθήσει να αποζητήσει μία συνένεση ή τουλάχιστον μία πλειοψηφία. Γιατί όπως βλέπω τα πράγματα εγώ, κυρία Γόλης, ε, όλοι έχουν σαφείς απόψεις, υπάρχουν αυτοί που τάσσονται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης, άλλοι ακολουθούν τη δική σας θέση περί επισήμανσης, άρα θα πρέπει να ψηφίσουν. Το αφήνω λοιπόν σε εσάς να το συζητήσετε με τους σκιώδεις και να δείτε κατά πόσο μπορείτε να φτάσετε σε μια συμφωνία. Θα ήταν πολύ καλό για την εικόνα αυτής της Επιτροπής να το επιλύσουμε κάπως από το να έχουμε μερικούς δυσαρεστημένους γιατί λαμβάνουμε σωρία email και από τις δύο πλευρές και θα προσπαθήσουμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τους ε, περισσότερους. Λοιπόν, προθεσμία θα ψηφίσουμε στις 2 Μαρτίου και έτσι έχετε αρκετό χρόνο να το συζητήσετε και με τις τροπολογίες επίπεδο να δείτε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ωραία, σας ευχαριστώ. Προτρέχουμε του χρόνου κατά 10 λεπτά. Θα μιλήσεις πάλι εξ ονόματος του Μάλκομ. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Έχουμε μεγάλη αποψήλωση από ό,τι βλέπω, αλλά εφόσον το ΕΛΚ είναι παρόν, μπορούμε να αρχίσουμε με τη συζήτησή μας. Θα Ήθελα να σας ενημερώσω ως προς τη διαδικασία που ε, εγκρίναμε για την οδηγία για τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θυμόσαστε ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόταση για τους ε, καταναλωτές με διτό στόχο να εξασφαλίσουμε στις επιχειρήσεις και τις μικρές ιδιαίτερα να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε 27 κράτη-μέλη με μία σειρά κανόνων, αλλά και οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη και υψηλό επίπεδο προστασίας κατά την πρόσβαση στις διασυνοριακές προσφορές. Συμφωνούμε με τους στόχους και αυτό που θέλουμε τώρα είναι να δούμε την πρόταση λεπτομερώς λήφθη μία απόφαση στους συντονιστές ότι θα δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας με επικεφαλής εμένα, με τον αντιπρόεδρο, τους συντονιστές όλων των πολιτικών ομάδων. Έχουμε κυρία Γόλης από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για ενισχυμένη συνεργασία και έχω λάβει και μία επιστολή από τον πρόεδρο τον κύριο Γκαργκάνη, που θα ασχοληθεί με το συμβατικό δίκαιο και το κοινό πεδίο αναφοράς το οποίο χρειαζόμαστε στα πλαίσια της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία εργασίας και υπάρχει και μια απόφαση η οποία ελήφθη από την ομάδα ε, εργασίας και από τις πολιτικές ομάδες κυρίως, διότι μέσα στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης θεώρησαν ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι επαρκές γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Το δέχομαι αυτό, γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία να μπούμε σε λεπτομεριακή εργασία, να έρθουμε σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς και να έχουμε μια καλή λειτουργική οδηγία και όχι να περάσουμε κάτι στα γρήγορα με ανεπίλητα ζητήματα. Άρα δεν θέλουμε μόνο ένα έγγραφο εργασίας, να συντάξουμε ένα έγγραφο εργασίας. Ε, το συζητήσαμε με την Επίτρεπο Κούνεβα για να καταλήξουμε σε μια προφορική ερώτηση με συζήτηση και ενδεχομένως ένα ψήφισμα για να αναγνωρίσουμε ορισμένα από τα θέματα που θίγουμε στο έγγραφο εργασίας. Έτσι έχει η διαδικασία η οποία ενεκρίθη. Φαντάζομαι ότι θα είδατε την ε, πρόταση. Ε, εδώ συγχωνεύονται αρκετές οδηγίες από την Πράσινη Βίβλο για τις πωλήσει πόρτα-πόρτα, για εξαποστάσεως συμβάσεις, συμβαστικό δίκαιο, εγγυήσεις μέσα στα πλαίσια της πλήρους εναρμόνισης. Και εδώ είχαμε εκπροσώπηση από πολλές οργανώσεις ανά την Ένωση. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα των κοινών ορισμών, του καταναλωτή, του εμπόρου, τι σημαίνει σύμβαση. Επίσης ε, συγκεκριμένες παραγγελίες από διαδίκτυο με φάξ ή δια τηλεφώνου και τι γίνεται πριν από τη σύναψη της ε, συμφωνίας αυτό το ξέρουμε και μέσα στα πλαίσια του δικαιώματος απόσυρσης, μέσα στα πλαίσια των 14 ημερών. Αυτό το είδαμε στην οδηγία χρονομερισμού, time share, και σε σχέση με τα, τους καταναλωτές, τα δικαιώματα καταναλωτών και τις υποχρώσεις του εμπόρου, ε, είναι υπόλογος για δύο χρόνια έναντι του καταναλωτή και σε άλλες χώρες ισχύουν διαφορετικά χρονικά περιθώρια μέσα στα πλαίσια του δικαίου υπέρ του καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ορισμένα ειδικά ζητήματα που εγκύπτουν. Και υπάρχει και το θέμα της νομικής ασφάλειας σε σχέση με τον καταναλωτή και τον έμπορο, τον επιχειρηματία. Σε μία συνάντηση είπαμε ότι θα ασχοληθούμε και με την ε, μελέτη αντικτύπου. Ένας συνάδελφος ε, μας έκανε μία παρουσίαση για την εκτίμηση αντικτύπου σε σχέση με την πρόταση που έχουμε επιτάπητος και ορισμένα ζήτημα εφήγησαν ως προς την εμβέλεια της οδηγίας. Δηλαδή σε σχέση με τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες για τι αποκλείονται από αυτή την οδηγία. Μας είπε η Επιτροπή ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συμπεριληφθούν αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης γιατί η εμβέλεια αφορά τις τέσσερις μόνο αυτές οδηγίες και η άποψη της Επιτροπής ε, ήταν ότι υπάρχει συνέργεια μεταξύ μόνο αυτών των τεσσάρων οδηγιών. Ο κύριος ε, Χάρμπορ μίλησε και για αυτορύθμιση και είπαμε ότι δεν αποκλείεται μπορούμε να την προσθέσουμε, αλλά χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο σε σχέση με την αυτορύθμιση για να προωθήσουμε το όλο πλαίσιο. Η κυρία Γκέπχαρτ αναρωτήθηκε πώς προβήκαμε στην επιλογή αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στοιχεία που έχουν εναρμονιστεί πλήρως και άλλα όχι. Αυτά είναι τα στοιχεία που ανακύπτουν. Και ένα άλλο σημείο που προώθησε η Επιτροπή ήταν το εξής. Είπαμε ότι στην μελέτη αντικτύπου θέλουμε να δούμε και θέματα συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αλλά οι καταναλωτές μας ερωτούν πώς αλλάζει η θέση τους ως καταναλωτές σε σχέση με την προσπελασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες στο κάθε κράτος μέλος. Και ξέρετε ότι αν εναρμονίζουμε, θα πρέπει να ξέρουμε σε τι επίπεδο εναρμονίζουμε. Υπάρχουν κράτη που έχουν άλλο κατόφλι, υψηλότερο ή κατώτερο. Και άλλοι καταναλωτές θεωρούν ότι χάνουν από αυτό το πλαίσιο, γιατί έχουν ανώτερο κατόφλι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η σημασία αυτών των αλλαγών και να δούμε κατά πόσο η Επιτροπή στη μελέτη αντικτύπου αναλύει αυτές τις αλλαγές. Λάβαμε σκόπιμες πληροφορίες. Η Επιτροπή έχει ένα συμπίλημα όλων των πληροφοριών από όλα τα κράτη-μέλη, άρα γνωρίζει τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Ζητήσαμε λοιπόν από την Επιτροπή να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πού επέρχονται αλλαγές ε, με βάση αυτή την οδηγία στους εθνικούς κανόνες. Δηλαδή αλλάζει το, αλλάζουν οι συμβάσεις, τα μέτρα αστικού δικαίου, τα μέτρα αποζημίωσης ή επανόρθωσης στα κράτη-μέλη ή δεν υφίσταται αλλαγή. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν οι αλλαγές που επέρχονται σε επίπεδο συμβατικού δικαίου και ε, ε, θα ήθελα λοιπόν να σας πω πώς έχουν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει αυτό το feedback. Εμείς πρέπει να παράξουμε ένα έγγραφο εργασίας. Στις 2 Μαρτίου θα γίνει μια δημόσια ακρόαση και θα καλέσουμε πολλούς ε, εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης θα προβάλλουμε και μία ε, διαβούλευση online καθώς και ένα κουτί όπου οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές θα μπορέσουν να μας δώσουν απαντήσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι, ποιος είναι ο βασικός στόχος, δηλαδή να ανοίξει η αγορά για όλες τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά και Παράλληλα, οι καταναλωτές να έχουν εγγυήσει για υψηλό επίπεδο προστασίας, δηλαδή να μην την χάνουν διακρίσεων έναντι αυτών των αγαθών και υπηρεσιών. Σας έδωσα μία... Ε, τη γενική εικόνα μάλλον της κατάστασης και θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε τα μέλη της ομάδας εργασίας και άλλα μέλη για το ποια είναι η άποψή τους, οι ανησυχίες τους και ούτω καθεξής. Ως προς τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε να σχολιάσετε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση στις πολιτικές <clears throat> ομάδες για να προωθήσουμε αυτή την εργασία και στην Ολομέλεια θα το προωθήσουμε ως προφορική ερώτηση ή προφορική ερώτηση με συζήτηση και ε, ψήφισμα. Ο κύριος Φάμπ, Φορτού και Ρούλε. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε ε, στο δύσκολο αυτό θέμα που μας μένει να εκπονήσουμε μέχρι τέλος της ε, κοινοβουλευτικής περίοδου. Στην ομάδα εργασίας, όπου συμμετέχει και ο Μάλκομ Χάρμπορ, αλλά σήμερα είναι απόν, έχουμε ήδη θέσει ορισμένα δύσκολα θέματα, τα οποία εσείς εξηγήσατε τώρα ε, ξεκάθαρα. Πάντως η συνεργασία μας είναι επικοδομητική. Ναι, μεν υπήρξαν στην αρχή κάποιες δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι από την εργασία μας θα προκύψει μια ακόμα καλύτερη πρόταση. Καταρχήν, εμείς σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Κομισιόν για το πεδίο εφαρμογής των τεσσάρων οδηγιών, θεωρούμε όντως ότι υπάρχει ανάγκη εναρμονίσεως μεταξύ των διαφόρων οδηγιών, αλλά πρέπει επίσης να κλείσουν ορισμένα κενά ανάμεσα στην εφαρμογή εθνικού δικαίου και βέβαια στην εφαρμογή κάποιες από τις οδηγίες, δηλαδή ε, ευρωπαϊκού δικαίου. Τώρα ελέγχθη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει κάποιες ε, ιδέες για το πώς θα μπορούν να συμβαδίζουν οι εφαρμογές των οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι είναι και θέμα λίγο ιδεολογικό για την ενιαία αγορά. Δηλαδή δεν αρκεί να βγαίνουμε μόνο να μιλούμε περί ενιαίας αγοράς ενώ όταν τίθεται θέμα εφαρμογής κάποιων πραγμάτων στην πράξη ε, να αποφεύγουμε. Από την άλλη μεριά βέβαια πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση και με κριτικό πνεύμα διότι βλέπουμε ότι σε ορισμένα σημεία τουλάχιστον έχει γίνει μια βιαστική επεξεργασία του κειμένου και δεν καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα. Βέβαια πρέπει να πω κιόλας ότι η Επιτροπή και η Συγκίδρια έχει αναλάβει υπερβολικό έργο διότι είναι πάνω από 20 ε, ένομες τάξεις διαφορετικές και είναι δύσκολο να τις συγκεράσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της ακροάσεως με ενδεχόμενο να καταθέσουμε πρόταση ψηφίσματος για την Ολομέλεια. Καταρχήν υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα όμως δεν γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι προσπάθειές μας για βελτίωση της προτάσεως αυτής. Και πάντως οι επικοδομητικές προτάσεις των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών μας ενδιαφέρουν δεν θέλουμε βέβαια να προωθήσουν μονάχα οι κυβερνήσεις τις δικές τους κάπως εγωκεντρικές ιδέες για τα συμφέροντά τους, αλλά να λάβουν υπόψη και τις απαιτήσει των άλλων μερών. Ωραία. Νομίζω πολύ επικοδομητικά τα όσα είπατε. Κυρία Φουρτού. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δύσκολο να προσθέσουμε πολλά περισσότερα από αυτά που είπε ο κύριος Υπάρχει κάτι το οποίο είναι λίγο παρακινδυνευμένο, δηλαδή εάν έχουμε έναν κατάλογο των διαφορών που υπάρχουν σε κάθε χώρα, παραδείγματος χάρη στην Γαλλία οι καταναλωτές ε, τη πολύ καλής μεταχείρισης. Εάν λοιπόν τότε αρχίσουμε να περιορίζουμε τα προνόμια μας και τα πλεονεκτήματα, τότε θα, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι τα προνόμια και να διατηρηθούν. Κύριε Φορτούρου, θα πρέπει πάντα κανείς να υπολογίσει τα υπέρ και τα κατά σε μια συζήτηση. Εμεί ε, θέλουμε να πετύχουμε μια εναρμόνιση και αυτό προς όφελος του καναλιού και της αγοράς. Κυρία Ρούλα. Ήθελα μετά την κυρία Φορτού να κάνω και εγώ μια σύντομη παρατήρηση. Στις χώρες μέλη πρέπει να πείσουμε και τα εθνικά μας κοινοβούλια. Άρα πρέπει να είναι απολύτως ενήμερα τα εθνικά κοινοβούλια για το τι σημαίνει η οδηγία. Ποια πράγματα θα βελτιωθούν και ποια θα επιδεινωθούν. Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι μεν έχει Κάποιε ιδέες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τι τοποθετήσει των ε, κυβερνήσεων, αλλά δεν αρκεί αυτό. Νομίζω ότι όλοι βέβαια θα χάσουν ή θα κερδίσουν κάτι όταν θα γίνει μια προσπάθεια συμβασμού, αλλά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και οι χώρες μέλη πρέπει και αυτές να προσεγγίσουν. Κύριε Βάιλερ, Σίγουρα θα πρόσθετα καταντελήφθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει εδώ συνένεση μεταξύ των Ευρωβουλευτών σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία. Άκουσα ω είπε ο αλλά ίσω δεν πρόσεξα καλά την πρώτη του ε, φράση. Δεν θέλουμε να υπάρξει πίεση χρόνου, διότι βεβαίω έχουμε τις ευρωεκλογέ και υπάρχει ο κίνδυνο να μα να το πω, στριμώξουν λίγο οι τα διάφορα συμφέροντα είναι πάρα πολύ έντονα. Το αποδεικνύει αυτό η τεράστια αλληλογραφία που λαμβάνουμε από διάφορες οργανώσεις. Είναι λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα σωστότερο, σκοπιμότερο και σημαντικότερο να τα αφήσουμε για μετά τις ευρωεκλογέ. Θεωρώ λοιπόν και από την άποψη αυτού του χρόνου πολύ σημαντικό αυτό. Ούτε είμαι βεβαία ότι αυτή η μία ακρόαση που προβλέπεται για αρχές Μαρτίου θα είναι αρκετή συμπτωματικά εγώ δεν μπορώ να είμαι παρούσα. Το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει όλους που ασχολούμαστε με θέματα προστασίας καταναλωτών. Ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί κάτι για το φθινόπωρο για παράδειγμα, για όλη την κοινοβουλευτική μας επιτροπή και ίσως οι πολιτικές ομάδες μπορούν να διεξαγάγουν κάποιες ακροάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να αντισταθούμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια πίεση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρονική πίεση δηλαδή. Ο κ. Σακελάκα. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο σχόλια γενικά. Επί της αρχής είναι καλοδεχούμενη κάθε προσπάθεια που εναρμονίζει την αγορά, βελτιώνει τις διασυνοριακές συναλλαγές, αλλά επειδή εδώ είμαστε η Επιτροπή των Καταναλωτών πρέπει να ενδιαφερόμεθα για το συμφέρον των καταναλωτών, γιατί αυτή είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής. Διαβάζοντας ε, την οδηγία, βλέπω ότι σε ορισμένα σημεία υπάρχει οπισθοδρόμηση, τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από συναδέλφους που μίλησαν, σε σχέση με τις διατάξεις που υπάρχουν σε εθνικά νομοθετικά πλαίσια. Ε, ενδεικτικά ζητήματα εγγυήσεων των, των αγαθών που αγοράζονται, ζητήματα εγγυήσεων των ανταλλακτικών συσκευών που αγοράζονται, ζητήματα όταν ένα αγαθό μεταβιβάζεται από τον ένα χρήστη στον άλλον ότι χάνεται η εγγύηση αυτά είναι θέματα που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση και χρήζουν ε, προσοχής και μελέτης. Συμφωνώ και εγώ να πάμε σιγά σιγά ε, ούτω ώστε να μην ε, παίξει μεγάλο ρόλο όσον αφορά την εκλογική διαδικασία διότι όλοι ξέρουμε ότι τα θέματα τα καταναλωτικά οι πολίτες θα παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή και έχουν απαιτήσει από εμάς ε, θεωρώ ότι όταν θα μπούμε στην ουσία της συζήτησης πολλά πράγματα θα ξεκαθαριστούν, αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχουν απορίες. Ευχαριστώ. Ε, Η κυρία Wallace, ε, ως εισηγήτρια από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, ζητώ συγγνώμη γιατί έπρεπε να βγω από την αίθουσα. Άρα δεν άκουσα όσα ελέγχθησαν στην αρχή της συζήτησης και λυπάμαι γιατί δεν ήμουνα και στην ομάδα εργασίες ε, σήμερα το πρωί και ήρθα από την Νορβηγία χωρίς βεβαίως να ασχολούμαι εκεί με ζήτηματα φώκιας. Δεν άκουσα λοιπόν την αρχή της συζήτησης, αλλά ελέγχθη αρχικά να μην γίνει η ακρόαση, γιατί από πλευράς Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την εργασία μας και ακόμα και σε αυτό το στάδιο πριν από τις ε, εκλογές να ακούσουμε την ε, άποψη των διαφόρων εμπειρογνωμόνων. Γι' αυτό θα πρότεινα να προχωρήσουμε με την προτινόμενη ακρόαση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική. Λοιπόν, η Επιτροπή θέλει το λόγο, καταρχήν, για να απαντήσει σε ορισμένα τα σχόλια που ακούστηκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από την σαφήνεια της ανάλυσής σας, ε, είμαι κάπως επιφυλακτικός ως προς το να λάβω το λόγο. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε εκτός από ένα σημείο διασάφησης στο τελευταίο σημείο που, που αναφέρατε. Πιστεύουμε ότι έχουν ακουστεί πολλές επικρίσεις από τις ενώσεις καταναλωτών για την πρόταση αυτή, γιατί δεν μπορέσαμε να αποστείλουμε αυτό το μήνυμα ε, αρκετά με αρκετή σαφήνεια από το κείμενο. Άρα υπάρχει η ερμηνεία του αντίκτυπου της πλήρους εναρμόνισης των εσωτερικών ενόμων τάξεων και αυτό εξηγούμε στον πίνακά μας, ένα συνοδευτικό συγκριτικό πίνακα. Εδώ στην αναθεώρηση του κεκτημένου ακολουθήσαμε μία προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή έχουμε εναρμονίσει πλήρως μόνο τα θέματα που καλύπτονται από τις υποαναθεώρηση οδηγίες, δηλαδή ως προς ε, θέματα ενοχικού δικαίου, τα οποία επεξημούνται στη μελέτη αντικτύπου, θέματα ενοχικού δικαίου, δηλαδή σύμβαση, σύνταξη, ε, σύνταξη της ε, συμφωνίας μετραποζημίωσης, ακυρότητα της σύμβασης, ε, δυνατότητα αποφυγής ε, της σύμβασης, όλα αυτά βρίσκονται εκτός εμβέλειας οδηγίας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα αυξήσουμε συνολικά το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και δεν θα μειώσουμε το εθνικό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Άρα η πλήρης εναρμόνιση των ε, κανόνων ως προς το συμβατικό δίκαιο υπέρ του καταναλωτή δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα ε, παραδοσιακά μέτρα ε, αντιστάθμισης ή αποζημίωσης με βάση το εθνικό ενοχικό δίκαιο. Αυτό θα το δούμε και στη συγκριτική ανάλυση, στο συνοδευτικό σημείωμα. Αυτά που είπε η κυρία Φορτού ε, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Γιατί είναι κάτι το σαφέστατο. Η πλήρης εναρμόνιση σχετίζεται με τα στοιχεία που εμπίπτουν στην εμβέλεια της οδηγίας, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αλλά θα έχουμε ορισμένες απώλειες αλλά ορισμένα και ορισμένα πλεονεκτήματα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ορισμένα κράτη-μέλη χάνουν σε μερικά σημεία και κερδίζουν σε άλλα. Αλλά το πιο σημαντικό μήνυμα Ε, στο οποίο προσδένεται και η μελέτη αντικτύπου σχετίζεται με το ότι έχουμε μια σχέση απολύτου κέρδους για τον ε, καταναλωτή, ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμμόρφωση, το κόστος συμμόρφωσης της επιχειρήσης και αυτό όχι σε περίπτωση διαφοράς, αλλά θα μειωθεί το συνολικό κόστος και θα υπάρχει νομική προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές έτσι ώστε ο δανός καταναλωτής που θεωρεί ότι έχει την καλύτερη δυνατή προστασία θα μπορέσει να εξάγει τα δικαιώματά του όταν μεταβεί στην Ιταλία και αγοράσει κάτι από την Ιταλία. Διότι τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή που εναρμονίζονται από αυτή την οδηγία θα είναι τα ίδια. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ίσως θα μπορούσα να σας πω ποια είναι η διαδικασία επί της οποίας έχουμε συμφωνήσει. Κυρία Βάιλερ, κατανοώ τις ανησυχίες σας, αλλά κάθε, δεν μπορούμε να λέμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές δεν θα ασχοληθούμε με ένα θέματα. Αυτό με κουράζει ιδιαίτερα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ψηφίσουμε επειδή έχουμε εκλογές. Θα πρέπει να επιτελεστεί αυτή η εργασία. Και δεν θέλουμε να το περάσουμε επειδή έχουμε εκλογές ή να μην το περάσουμε, αλλά θεωρούμε ότι είναι περίπλοκο ζήτημα. Θα πρέπει να μας απασχολήσει για να το πετύχουμε και για να ικανοποιήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε είναι επιχειρηματίες είτε είναι καταναλωτές. Δεχόμαστε τους στόχους ε, της οδηγίας να ανοίξει δηλαδή η εσωτερική αγορά με μία σειρά ενιαίων κανόνων, αλλά θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να μην ζημιωθεί ο καταναλωτής σε σχέση και με την εθνική νομοθεσία. Δηλαδή δεν θα ισχύσει το διέρη και βασίλευε, θα δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα σε κάθε κράτος μέλος, διότι έμπρακτα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα γίνει ακρόαση στις 2 Μαρτίου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν θα έχουμε πρώτη ανάγνωση τροπολογία σε αυτό το στάδιο. Θα έχουμε και μία διαβούλευση online με μία σειρά ερωτημάτων που έδωσα στην ομάδα εργασίας για να προσθέσουν ή να τροποποιήσουν ενδεχομένως έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μας κοινοποιήσουν όχι μόνο τις απόψεις τους, μερικοί είναι σύμφωνοι, άλλοι όχι, αλλά θα θέλαμε και ιδέες ή εναλλακτικές εάν υπάρχουν για την επίτευξη των στόχων. Και όπως σας είπα, Συμφωνήσαμε ήδη ότι θα έχουμε ένα έγγραφο εργασίας και μετά θα έχουμε σύνταξη μιας προφορικής ερώτησης, ενδεχομένως με ψήφισμα και μια συζήτηση με την Επίτροπο. Θα δούμε κατά πόσο θα είμαστε θέση να συντάξουμε και ψήφισμα, το οποίο θα είναι μια πολύ καλή κληρονομιά για το επόμενο Κοινοβούλιο δεν ε, σημαίνει ότι επειδή την ε, πρόταση τη λάβουμε τον Οκτώβριο του 2008 δεν μπορούμε να την προωθήσουμε. Και το επόμενο κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο και μπορεί να αποφασίσει να δεχτεί ή όχι την πρόταση. Θα αφήσουμε λοιπόν αυτή την κληρονομιά για να πληροφορήσουμε το επόμενο κοινοβούλιο. Και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με αυτή την απόφασή μας. Η κυρία Γουόλης... Η κυρία ξέρετε ότι θα λάβουμε υπόψη και θέματα που αφορούν την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Υπάρχει ένα τρίτο τμήμα στην ακρόαση που αφορά τους κοινού όρους αναφοράς και το ενοχικό δίκαιο και πολλοί καθηγητές θα λάβουν το λόγο, αλλά η κυρία Γουόλης θα αποφασίσει τι θέλει να λάβει υπόψη σε αυτό το τμήμα της ακρόασης γιατί υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία σε αυτό το τομέα. Άρα βασίζομαι σε εσάς να ασχοληθείτε με τα θέματα που κρίνετε σημαντικά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Θα ήθελα την υποστήριξη της Επιτροπής έτσι ώστε να ασχοληθούμε με τις πρακτικές πτυχές του ζητήματος, γιατί πρέπει να δώσουμε μία απάντηση στους εμπλεκόμενους φορείς δηλαδή γιατί δεχόμαστε ορισμένες προτάσεις Επιτροπής, γιατί ε, πρέπει να επέλθουν αλλαγές σε άλλους τομείς και αυτό είναι και το πλέον λογικό που μπορεί να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα και το γεγονός ότι σχεδόν λίγη η θητεία μας. Δεν έχω άλλα να αναφέρω γιατί σας είπα, σύντομα θα γίνει η ακρόαση, θα έχουμε και μία ε, online διαβούλευση. Άρα θα έχουμε πολλές απόψεις που μπορούμε να ενσωματώσουμε στο έγγραφο εργασίας που θα προετοιμάσει η Γραμματεία ε, εξ ονόματος Ομάδας Εργασίας. Και θα ξαναγίνει η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή για να παρέμβουν και τα μέλη μπορούμε να λάβουμε υπόψη και μεμονωμένα σχόλια από τα μέλη που έχουν ειδικά ζητήματα για να τα δούμε εξ αρχής και όχι εκ των υστέρων. Αν δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα ή παρεμβάσεις, δεν ξέρω κατά πόσο το Συμβούλιο θέλει να λάβει το λόγο, όχι δεν υπάρχει και κανένας εκπρόσωπος από το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο προχωρά αργά επί του θέματος. Θέλετε να επανέλθετε επί του θέματος. Η κυρία Βάιλερ, σύντομη ερώτηση. Μετά την ακρόαση θα συνταχθεί working document και μετά το χρονοδιάγραμμα ποιο θα είναι περίπου. Πρόεδρος, θα εργαστούμε διαδοχικά στην ομάδα εργασίας και στην ακρόαση για να παραγάγουμε, για να συντάξουμε το ε, έγγραφο εργασίας που η προθεσμία είναι μέχρι τις 3 Μαρτίου. Και είπα επίσης ότι συμφωνώ, συμφώνησα με τον πρόεδρο Γκαργκάνη που δεν είναι νομίζω και θέμα, διότι και η κυρία Γόρης είναι μέλος και της παρούσης Επιτροπής, για να εργαστούμε χέρι με χέρι με την ε, νομική επιτροπή, να λάβουμε υπόψη και τις δικές τους θέσεις. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Είμαστε αρκετά μπροστά, συνήθως καθυστερούμε. Αλλά επειδή δεν είχαμε έντονη παρουσία μελών, προχωρούμε γρήγορα. Θα ήθελα τώρα, επειδή η κυρία Μπαρνιέ είναι εδώ, να εξετάσουμε ορισμένες από τις τροπολογίες για τα δικαιώματα των ασθενών σε διαμεθοριακές φροντίδες υγείας. Πάντως, δεν αντιμετωπίζουμε τον ίδιο επίγοντα χαρακτήρα διότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει αναβάλει την ψηφοφορία της. Είμαι βεβαίω ότι θα μπορέσετε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Και έχουμε και αίτηση προς την νομική επιτροπή για να κάνει μια νομική γνωμοδότηση για, την, ε, για το θέμα αυτό. Άρα δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να επιταχύνουμε πάρα πολύ τις διαδικασίες και τις ψηφοφορίες. Μου είπαν επίσης οι συντονιστές να σας πω να επανέλθω στο θέμα με τον κύριο Ούσκι. Δεν έχουμε ακόμα δηλαδή συμφωνία για θέματα αρμοδιοτήτων. Διότι ε, σύμφωνα με το άρθρο 47 είμαστε σε ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή του και με τον κύριο Γαλεώτε που είναι ο πρόεδρος των προέδρων των ε, ε, Επιτροπών και με τον κύριο Ούσκι συζητούμε εν πάση περιπτώσει ώστε να τα βρούμε. Κύριε Ενιούλ, να σας δώσω το λόγο για να μας τα πείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα με τα νέα που μόλις μας ε, είπατε, διότι πηγαίνουμε στην κατεύθυνση των ετοιμάτων της Επιτροπής μας. Λοιπόν, αν υπάρξει μετάθεση της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ήταν καλό, διότι έμαθα σήμερα πως ε, και στην Επιτροπή απασχόληση, η οποία πρόκειται να ψηφίσει σήμερα το πρωί τελικά δεν ψήφισε και πω η Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, έπραξε το αυτό. Όντω παραμένουν τα προβλήματα τα οποία δεν ρυθμίστηκαν ακόμα, δηλαδή προβλήματα αρμοδιότητα. Και αναθέσαμε στην νομική υπηρεσία να το εξετάσει και μα είπε ότι θα μα προφορήσει την 3η Μαρτίου. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε στις 2 Μαρτίου, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να μεταθέσουμε την ψηφοφορία μας. Θεωρώ πως οι συντονιστές και οι πρόεδροι των εμπλεκομένων επιτροπών θα ορίσουν την ημερομηνία και θα μας την ε, ανακοινώσουν. Έχω κάποια άλλα προβλήματα να σας ε, θέσω και είναι φυσιολογικό. Είναι ένα φάκελο ιδιαίτερα περίπλοκο. Ε, όταν είπα πω θα χρειαστούμε χρόνο, Υπάρχουν 27 κρατη 27 διαφορετικά συστήματα υγείας. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το ζήτημα, με πάρα πολλές τροπολογίες, 371 συγκεκριμένα από όλες τις πολιτικές ομάδες. Το μόνο πρόβλημα το να ζητηθούν σήμερα είναι πως μέχρι τούδε δεν έχουμε λάβει καμία μεταφρασμένη τροπολογία. Εγώ μπορώ να εξετάσω τις γαλλικές και τις ισπανικές τροπολογίες, αλλά τις υπόλοιπες δεν είναι δυνατόν. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πως σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά, επιχειρηματολογώντας, δίχως να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των τροπολογιών. Βλέπω παραδείγματος χάρη πως ε, η κυρία Ρόιτοβα, η κυρία Σέντε ε, η κυρία Τίσεν, που και αυτή έχει καρθές πολλές τροπολογίες, η κυρία Μπέργκερ, ε, η Μάρτη επίσης, απουσιάζουν, μόνο η κυρία Ρόιτοβα είναι παρούσα και μια που δεν υπάρχει μετάφραση θα πρέπει να βρούμε κάποια άλλη ημερομηνία για να τις εξετάσουμε τις τροπολογίες αυτές. Και για να διευκολύνω τις εργασίες μας πιστεύω πως η μετάφραση θα είναι έτοιμη σε μια-δυο μέρες και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε όλοι οι σκιώδεις την προσεχή εβδομάδα αν έχετε δυνατότητα στην 5η 19 το πρωί, διότι είναι η μήνυ ολομέλεια στις Βρυξέλλες, το πρωί της 5ης 9 με 10, πριν από την έναρξη της ε, ολομέλειας, ε, στην οποία θα παραστεί και η Τσεχική Προεδρία, θα είναι η πανηγυρική. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, περιμένουμε κυρία Πρόεδρε το θέμα της νομικής βάσης. Ε, βρίσκεται σε εξέλιξη το θέμα. Έχουμε επίση το, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν έχει ακόμα επιληθεί και ίσω χρειαστεί να το συζητήσουμε όταν θα γνωρίσουμε όλε τις τροπολογίε. Για μένα τα θέματα που θέτει το άρθρο 5, δηλαδή την ευθύνη των κρατών μελών, Ορισμένοι λένε πώ δεν υπάρχει οι δυσκολία σε επίπεδο συμβουλίου, διότι τα κράτη-μέλη φαίνεται πώ συμφωνούν. Ε, εγώ έχω άλλε ειδήσει, τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν και θα πρέπει να το εξετάσουμε και συνδέεται εδώ με το 5 το άρθρο 11 που αφορά την ε, θεραπεία το δικαίωμα του κράτους ε, ασφάλισης ή το, το δίκαιο του κράτους ασφάλισης ή το δίκαιο του κράτους ε, νοσηλείας θα πρέπει λοιπόν επίσης να βρούμε και το θέμα του ορισμού των νοσοκομιακών ε, της δοξοσιομικής φροντίδας λοιπά. Επαναλαμβάνω λοιπόν την πρότασή μου, διότι θεωρώ πως σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε μεταφρασμένες τροπολογίες. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πολύ λεπτό. Κυρία Ρόιτοβα, έχετε καταθέσει πολλέ τροπολογίε. Θα ήθελα να τι διαβάσω, αλλά δεν καταλαβαίνω μία από την γλώσσα σα και ούτε και τη γλώσσα της κυρία Τάισεν. Ας ε, ακούσουμε τους Κιώδης. Κύριος Φαμπ. Ναι, δεν λέγομαι Μποκ, μα δεν νομίζω ότι του μοιάζεται κιόλα. Αλλά ο κύριος Μποκ είπε ότι έρθει στις 5, δεν ξέρω αν θα φτάσει έγκαιρα. Θα προσπαθήσω πάντως, όσο μπορώ τουλάχιστον, να αναπτύξω ορισμένα θέματα της απόψεως του ΕΛΚ ε, για την εργασία της κυρίας Μπρινιό. Πρώτα, νομίζω ότι πρέπει όντως να ολοκληρώσουμε την εργασία που έχει ήδη αρχίσει. Και τα διάφορα παιχνιδάκια τα οποία παίζουν διάφορες πλευρές με πραγματογνωμοσύνες οι οποίες εμφανίζονται ή υποτίθεται θα εμφανιστούν μια μέρα μετά από τις ψηφοφορίες που γίνονται σε διάφορες άλλες επιτροπές αυτά τα παιχνιδάκια νομίζω είναι άσκοπα, διότι πρόκειται για ένα θέμα θεμελιώδες για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το μεγάλο πλήθος των τροπολογιών, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του φακέλου. και να καταλήξουμε στη συμφωνία ήδη μέσα στα πλαίσια τη παρούσα κοινοβουλευτική περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, για τη δική μα πολιτική ομάδα είναι σαφέ ότι πρέπει να αναζητήσουμε την μέση οδό μεταξύ των συμφερόντων των χωρών μελών από τη μια μεριά, οι οποίε για διαφόρου λόγου έχουν προβλήματα με τα συστήματα υγεία του. Για παράδειγμα, ορισμένε έχουν πολύ περιορισμένο προσωπικό εκπαιδευμένο και είναι αναγκασμένες να προσπαθούν να προσλάβουν προσωπικό είτε από άλλες χώρες μέλη είτε από τρίτες χώρες για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα υγείας τους. Άλλο ε, πρόβλημα είναι των συστημάτων υγείας τα οποία δαπανούν πολλά ωστόσο προσφέρουν περιορισμένες ή κακής ποιότητας υπηρεσίας. υπηρεσίες. Είναι βεβαίως αυτά θέματα αρμοδιότητας των χωρών μελών. Από την άλλη μεριά θεωρώ πάντως ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παρούσα οδηγία ώστε να μειώσουμε τα δικαιώματα τα οποία έχει ήδη αναγνωρίσει με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπέρ των Ευρωπαίων ασθενών. Θεωρώ ότι βέβαια βρισκόμαστε και ενώπιον ευρωεκλογών και έχουμε και την έξτρα δυσκολία να πείσουμε τους εθνικούς βουλευτές συναδέλφου μας και να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο θεωρούμε ότι έχουν προτεραιότητα τα δικαιώματα των ασθενών απέναντι στα συμφέροντα των χωρών μελών. Εγώ θεωρώ πάντως ότι ως Επιτροπή Ενίας Αγοράς δεν έχουμε και καμία εναλλακτική επιλογή. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προωθήσουμε την διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει με την καθοδήγηση της ε, εισηγητρίας κ. Μπερνιό να καταλήξουμε σε στέρεες συμφωνίες και συμβιβασμού ώστε τελικά να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και σε αυτά που έχει ήδη αναγνωρίσει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δηλαδή τα δικαιώματα των ασθενών. Όπως γνωρίζετε, 1% μόνο των χορηγουμένων φροντίδων υγείας καλύπτεται από την παρουσία οδηγία. Είναι δηλαδή διαμεθοριακού χαρακτήρα που εμπίπτει σε αυτή την οδηγία. Αυτό το 1% λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίζει την ίδια, τον ίδιο καταμερισμό και την ίδια παροχή δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την κοινωνική διαστρωμάτωση των ασθενών που υποφελούνται από, τα, από τις φροντίδες αυτές, όπως και το υπόλοιπο 99%. Ευχαριστώ. Κύριε Ρίς Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Περνό, συμφωνώ μαζί της ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα διότι δεν έχουμε τις μεταφράσεις. Εγώ καταλαβαίνω πολλές γλώσσες αλλά δεν καταλαβαίνω τα φλαμανδικά. Δεν μπορώ λοιπόν να διαβάσω τις τροπολογίες της κυρίας Τάισεν. Με δυσαρεστεί λίγο το γεγονός διότι περνούμε χρόνο εδώ για να παραλαμβάνουμε πράγματα τα οποία έχουμε ήδη πει. Και όταν πάμε να μπούμε σε λεπτομέρειε, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Ενώ θα μα διευκόλυνε για να καταλήξουμε σε συνένεση. Δεν έχουμε τι μεταφράσει, όπω είπα. Δεν θα επαναλάβω τα όσα έχω πει παλαιότερα στι τροπολογίε μου. Δεν μπορείτε κι εσεί να τι διαβάσετε πριν να μεταφραστούν. Πάντως ελπίζω να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ένα χρονοδιάγραμμα τέτοιο που να μας επιτρέψει να ψηφίσουμε πριν από τις εκλογές. Και φοβούμε ότι πολλοί θα προσπαθήσουν να το βγάλουν το θέμα από την ατζέντα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε. Ίσως μπορούμε να αναβάλουμε για μία εβδομάδα, αλλά όχι περισσότερο παρακαλώ, διότι μας χρειάζεται αυτό το σημαντικό νομοθέτημα να ψηφιστεί δηλαδή πριν να φτάσουμε στις εκλογές. Η κυρία είναι ακούσα; Η κυρία Ρόιτοβα. Ε, Ευχαριστώ. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να συζητήσουμε διότι έχουμε στη διάθεσή μας ε, διερμηνία και θα ήθελα να επικεντρωθώ με ορισμένες που αφορούν ακριβώς ε, την αποσαφήνιση του κανόνα που θα έπρεπε να εφαρμόζεται για τους ε, ασθενείς οι οποίοι πριν να ζητήσουν τις να προσφύγουν στη θεραπεία πρέπει να ζητήσουν την άδεια και την ενημέρωση από την ασφάλειά τους ε, είναι γεγονό ότι οι τροπολογίε δεν είναι μεταφρασμένες αλλά υπάρχει μια κοινή βάση ότι δηλαδή το δικαστήριο έχει δηλώσει ότι δεν θα πρέπει <clears throat> να νοσηλεύεται χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη και αν η νοσηλεία αυτή είναι ιδιαίτερα δαπανηρή τότε εκεί είναι απαραίτητο ο ασθενής προηγούμενο να έρθει σε επαφή με το υγειονομικό σύστημα με την ασφάλειά του για να γνωρίζει τι θα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο ώστε να συμπεριλάβουμε μια διάταξη στην ε, οδηγία για το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να καθορίζεται κάποιος σαφής ε, κανόνας στην περίπτωση στην οποία ο ασθενής ε, δεν θα πρέπει να νοσηλεύεται δίχως την άδεια του του ασφαλιστικού φορέα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η νοσηλεία σημαίνει όταν υπάρχει διανυκτέρευση στο νοσοκομείο τουλάχιστον μιας νύχτας. Και εγώ θα ήθελα να διαγραφεί ο όρος εξειδικευμένες ε, θεραπείες. Εγώ θα ήθελα να αναφέρουμε τις ιδιαίτερα δαπανηρές ε, θεραπείες. Πρόκειται λοιπόν για θεραπείες οι οποίες κοστίζουν πάρα πολύ και το κόστος θα πρέπει να το κρίνει ο οργανισμός ασφάλισης και να εξεταστεί το κατά πόσον είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδα και σε κάθε χώρα θα πρέπει να υπάρχουν κατάλογοι για αυτούς, αυτές τις εξηγευμένες θεραπείες διότι πολύ καλά ότι η ιατρική εξελίσσεται συνεχώ και τουλάχιστον στη χώρα μου ε, έχω μια εμπειρία ότι οι γιατροί δύσκολα συμφωνούν. Άρα λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν κάποιο ανώτατο όριο δαπανών με το οποίο θα συμφωνούν και οι ιατροί αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Να υπάρχει λοιπόν κάποιο ανώτατο όριο και όταν οι δαπάνες που συνδέονται με συγκεκριμένη θεραπεία ξεπερνούν αυτό το ανώτατο όριο, αυτό θα είναι ένα δείγμα για τον ασθενή ο οποίος θα πρέπει να ταρθεί προς την ασφαλιστική του εταιρεία. Ω εκ τούτου λοιπόν δεν χρειάζεται να υπάρχει συγκεκριμένο ορισμός των εξειδικευμένων ε, θεραπείων Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι γνώμες διήστανται, δεν είναι κάτι το απλό, αλλά τα κράτη-μέλη μπορούν να προσδιορίσουν το ανώτατο όριο δαπάνης, σύμφωνα με το οποίο θα υποχρεούται ο ασφαλισμένος να απευθύνεται και να στανοείται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Νομίζω ότι η Κομισιόν εδώ θα πρέπει να παίξει τον ρόλο της και να διασφαλιστεί ότι αυτό το ανώτατο όριο είναι το πρέπον όπως έχει καθοριστεί από τα κράτη-μέλη αλλά είναι γεγονός ότι σε κάποιες χώρες θα είναι χαμηλότερο και σε άλλες υψηλότερο. Π.χ. υψηλότερο Ρουμανία, ε, Βουλγαρία θα είναι χαμηλότερο, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία θα είναι υψηλότερο. Επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα. Είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκα επισταμένος και αφορά την τόσο περίπλοκη πρόταση σε ό,τι την ανάγνωσή της τουλάχιστον είναι η πρόταση της κυρίας Βερνιού για την περαιτέρω απλούστευση του κειμένου αλλά στην έκθεσή της διαγράφει τις αναφορές που γίνονται σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα πρέπει να τηρήσουμε την οδηγία 1381 η Κομισιόν είναι, η ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την θέση της παρά μόνο εάν επαρθμίσουμε όλες τις περιπτώσεις όπου ο ασθενής θα, θα τηρεί την ε, κανονισμό 1381 ή και αν αυτός και αυτή η αναφορά στον νόμο κανονισμό δεν συμπεριλαμβάνεται. Πρόκειται για έναν εκτελεστικό κανονισμό. Κατά την άποψή μου λοιπόν η θέση της Επιτροπής είναι ορθή. Έχω και άλλες τροπολογίες, αλλά αυτές οι δύο θεωρώ ότι είναι σημαντικές και αν θέλετε μπορούμε να τις εξετάσουμε περαιτέρω και να φροντίσουμε να επιτύχουμε κάποια συνένεση αυτών. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έλθω. Με καθυστέρησε μια σημαντική συζήτηση που είχα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Το σύστημα είναι δύσκολο και περίπλοκο. Έχουμε πολλές τροπολογίες και μόνο στην Επιτροπή μας, οι οποίες δεν έχουν μεταφραστεί ακόμη. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, έχετε δίκιο, να συζητήσουμε σε βάθος. Θα χρειαστεί λοιπόν να προβλέψουμε νέες συζητήσεις. Και αυτό μάλιστα το έγγραφο που είναι αναμεμειγνύες τροπολογίες σε διάφορες γλώσσες μόλις τώρα το έλαβα. Και η συγκίτρια βεβαίω αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε λοιπόν. Θα αναφερθώ και σε ένα θέμα το οποίο έθεσα εγώ και επειδή βέβαια είναι νούμερα τα καταλαβαίνω χωρίς ιδιαίτερες γλωσσικές γνώσεις. Πρόκειται για το θέμα της νομικής βάσης. Σε ποια νομική βάση θα βασίσουμε την πρότασή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και όλοι μας είπαμε ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες για να προσεγγίσει κανείς το θέμα. Είτε πολύ στενά, ώστε να συζητήσουμε μόνο περί κινητικότητας των ασθενών, ώστε τότε το, 95, το 95 δεν μπορεί να είναι η σωστή νομική βάση, αλλά πρέπει να επιλεχθεί το 152 που αναφέρεται σε θέματα φροντίδας υγείας. Στην πρώτη μου θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουν μέρος της Νομικής Επιτροπής και εκεί αρμόδια για τις νομικές βάσεις. Και στις συζητήσεις έμαθα, εν πάση περιπτώσει, ότι προηγείται πάντοτε το ειδικότερο δίκαιο, το λέξη specialis. Όταν υπάρχει λοιπόν μια ειδική διάταξη, εφαρμόζεται αυτή και οι γενικότερες διατάξεις έρχονται και ισχύουν μετά από αυτήν. Εάν λοιπόν τελικώς συμφωνήσουμε ότι μας απασχολεί μόνο η κινητικότητα των ασθενών, τότε πρέπει να επιλέξουμε το άρθρο 152 ως νομική βάση. Είτε όμως και αυτή είναι η δική μου προτίμηση και εν των συζητήσεων που κάναμε για την ε, οδηγία περί υπηρεσιών να κάνουμε ένα συνολικότερο κείμενο ώστε τότε θα είναι το σωστό το άρθρο 95 αλλά θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό το σχέδιο που θα πρέπει να μας υποβληθεί το οποίο να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αξιώσεις δεν συνέβη κάτι τέτοιο βλέπω τώρα ότι ένας αριθμός συναδέλφων έχουν υποβάλει διαφορετικά πράγματα. Βλέπω 95, 16, 42, 308, διάφορα λοιπόν άρθρα, 137. Πολλές νομικές βάσεις οι οποίες έχουν προταθεί. Χθες ως συντονίστρια έμαθα ότι η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αυτή του περιβάλλοντος έχει ζητήσει από την νομική επιτροπή να εξετάσει ποια είναι η σωστή νομική βάση. Ρωτά όμως εάν η σωστή είναι η 95 ή 152 ή ένα συνδυασμό των δύο. Σωστό θα είναι η δική μας επιτροπή εν ώψη των πολλών προτάσεων νομικών βάσεων που κατατίθεται να ζητήσει και αυτή με ερώτησή της προς την νομική επιτροπή να μάθει τι πιστεύει η νομική επιτροπή για τις νομικές αυτές βάσεις. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει ζητήσει από την Γιούρη να ε, υποβάλει την γνωμοδότησή της μέχρι τις 3 Μαρτίου και εμείς έχουμε ορίσει ψηφοφορία στις 2 Μαρτίου. Θα προτείνω λοιπόν να αναβάλουμε την ψηφοφορία μας ώστε να έχουμε απαντήσει τις ερωτήσεις μας και να έχουμε μια καλή βάση για την ψηφοφορία. Δεν έχει νόημα εμείς να ψάχνουμε από εδώ και από εκεί μέσα στις συνθήκες να βρούμε την νομική βάση, τη σωστή νομική βάση. Είναι σωστό να μπορέσουμε να βασιστούμε σε μια νομική γνωμοδότηση. Αυτά για το θέμα αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και χθε άλλωστε το είπαμε μεταξύ των συντονιστών ότι πρέπει να το ε, εξετάσουμε. Το αίτημά μου τώρα για το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας και χωρίς να γνωρίζω τι περιέχεται στις 400 τροπολογίες είναι να κάνουμε πράγματι αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα κάνει. Να αναφερθεί δηλαδή μοναχά σε θέματα κινητικότητας των ασθενών και να διαγραφούν από την οδηγία όλα τα άλλα θέματα που έχουν σχέση δηλαδή με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών που έχουν ρυθμιστεί με την αμοιβή αναγνώριση τίτλων σπουδών κλπ. Είναι υπηρεσίε οι οποίε είναι ρυθμισμένε και υπηρεσίε υγεία μεταξύ αυτών και η ελευθερία εγκαταστάσεως και προσφοράς υπηρεσιών. Και νομίζω θα πρέπει να περιοριστούμε στο θέμα αυτό της κινητικότητας των ασθενών και να δούμε πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα δικαιώματα που διαθέτουν και τα οποία έχουν αναγνωριστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Χωρίς να διατρέξουμε και κίνδυνο τα συστήματά μας των χωρών μελών δηλαδή να αμφισβητηθούν. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Αφού πρέπει να είναι σαφές ένα πράγμα. Εφόσον τώρα ψηφίσουμε ένα νόμο εδώ και έχουμε συστήματα υγείας στις χώρες μας τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίε λόγω των δημογραφικών εξελίξεων. Και αν πρέπει να το λάβουμε αυτά υπόψη και να λάβουμε επίση υπόψη ότι οι υπηρεσίε που ε, προσφέρουν, που εξασφαλίζει η οδηγία παροχή υπηρεσιών υγεία είναι καθολικού χαρακτήρα. Άρα πρέπει να μπορούν να προσφέρονται παντού και σε υψηλή ε, ε, επίπεδο, επίπεδο ποιότητας. Διότι δεν θα μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε να κάνουν αυτά που λέει στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σηκωθούν να πάνε δηλαδή σε μια άλλη χώρα και να δεχθούν εκεί φροντίδε υγεία. και μάλιστα να μπορέσουν να δώσουν και τις απαραίτητες προκαταβολές και να επιστρέψουν μετά στις πατρίδε τους και να ζητήσουν επιστροφή των δαπανών του. Δεν μπορούν να κάνουν όλα, όλα όλοι οι πολίτε αυτά τα πράγματα. Μόνο αυτοί που είναι εύποροι μπορούν. Άρα πρέπει οι φροντίδες υγείας να χορηγούνται επιτόπου. Να παρέχονται επιτόπου. Αυτό είναι σαφές. Και συμφωνώ μαζί σας κυρία Ρόιτοβα. Όπως και να το κάνουμε. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Θα δούμε ποιες προτάσεις έχουν κατατεθεί, πώς μπορούμε να το εξασφαλίσουμε και να προπαρασκευάσουμε τη λήψη μιας σωστής αποφάσεως. Για την κυρία Γιώργενσεν Έχω ένα σχόλιο. Δεν θέλω να δεσμευτώ σήμερα για το πότε θα κάνουμε την ψηφοφορία. Και γνωρίζω ότι έχουμε διάσταση απόψεων. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει με κάθε προσπάθεια να κάνουμε ψηφοφορία στην επόμενη, επόμενο μήνα και μάλιστα σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς να γνωρίζουμε σαφώς τις συνέπειες, τις επιπτώσεις των όσων αποφασίζουμε εδώ, των όσων εδώ. Αν είναι δυνατόν, έχει καλώς αν είναι δυνατόν λέω, έχει καλώς, Αλλά όχι όμως να προαποφασίσουμε εκ των προτέρων ότι οπωσδήποτε θα το πράξουμε. Διότι εδώ πρόκειται για την υγεία των πολιτών, για τα δικαιώματα των ασθενών, για την προστασία των ασθενών. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε προσεκτικότατα το τι πράττουμε και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας. Δεν μπορώ να δεχτώ τίποτε άλλο από αυτά. Αν γίνεται λοιπόν έχει καλό, αλλά όχι να πούμε από την αρχή ότι πρέπει οπωσδήποτε να ψηφίσουμε, διότι τότε τα πράγματα θα πάνε άσχημα και τότε οι πολίτες θα γυρίσουν και θα μας πούν τέτοια Ευρώπη δεν την θέλουμε. Θέλουμε Ευρώπη υπέρ των πολιτών. Νομίζω Λέω, ο ότι αυτές οι προφυλάξεις είναι ουσιώδεις. Τα δικαιώματα των ασθενών είναι ύψης της σημασίας για την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις στα εθνικά συστήματα υγείας και στις εθνικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και τα εθνικά συστήματα ασφάλισης. Και αυτό αν δεν γίνει με μεγάλη προσοχή διατρέχουμε μεγάλους κινδύνους. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στην κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος και του ιατρικού συστήματος, του εθνικού συστήματος υγείας. Όπως είδατε, το αμερικανικό, η αμερικανική κρίση μόλυνε και την Ευρώπη και έτσι η οικοδόμηση των εθνικών συστημάτων υγείας θα καταρακωθεί εάν δεν ακολουθήσουμε μία εύλογη διαδικασία έρευνας. Θα καταρρεύσουν τα συστήματα και θα καταρρεύσουν και τα εθνικά συστήματα ασφάλισης. Αυτό το είδαμε και στην οδηγία περί όπως είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας και θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί. Εγώ έχω εργαστεί στο σύστημα εθνικής ασφάλισης και συμμετείχα και στην Επιτροπή, ε, Εθνική Επιτροπή Υγείας στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διαφορετικά κινδυνεύουμε με την κατάρρευση του συστήματος. Θα ήθελα όμως να συγχαρώ την κυρία Βερνιό. Η κυρία Ρίς και η κυρία Ρόιτοβα στη συνέχεια. Η κυρία Γιόργενσεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτή τη νομική βάση Κατανοώ ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ζήτησε ένα έγγραφο για να συζητήσει τη νομική βάση. Και ίσως δεν κατάλαβα τι είπε η κυρία Γκέπχαρτ, αλλά δεν χρειάζεται να το ζητήσουμε άλλη μια φορά. Αν υπάρχει αυτό το έγγραφο, καλώς. Δεν χρειαζόμαστε ε, έγγραφα νομικού περιεχομένου κανόνες, ε, ο κανονισμός ε, λέει ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα αποφανθεί. Αλλά η κυρία Γκέπχαρτ μίλησε για μία έκθεση και θα δούμε ποια, είναι, ποια θα είναι η έκβαση. Ωραία, τότε αυτό έχει διευθετηθεί. Χαίρομαι που είπε η κυρία Γκέπχαρτ ότι με βάση τις δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τήρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Υπάρχουν και πολλές τροπολογίες και στο τέλος λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία ή θα πρέπει να είναι μια εξαίρεση, να αποτελεί εξαίρεση. Ποιος τα θέλει όλα αυτά στην Ευρώπη. Οι πολίτες βέβαια θέλουν ιατρική περίθαλψη. Και όταν άκουσα τον συντονιστή της σοσιαλιστικής ομάδας, είναι σαν να μας λέει ότι αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την οδηγία, αυτό θα ήταν εξαιρετικό, διότι θα δημιουργήσει προβλήματα στα κράτη-μέλη. Βλέπω ότι όλοι αντιτάσσονται, αλλά αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση. Ας είμαστε ανοιχτοί και ας πούμε τι θέλουμε παρά να μιλάμε για φανταστικά ε, επινοήματα και στο τέλος να τα αποποιούμαστε. Κυρία ε, Ρόιτοβα, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο κύριος Χάσε Κύριε Φερέιρα, μπορείτε να καθίσετε εφόσον σε, σένα, σε εσάς απευθύνεται η ομιλήτρια. Τουλάχιστον καθίστε μέχρι να τελειώσει η παρέμβασή της. <laughs> Eh, eh, eh, Θα μιλήσω τσεχικά, κατανοώ αυτές τις ανησυχίες ότι διανύουμε μια περίοδο κρίσης και έτσι μπορεί να πλήξει τα συστήματα και αυτή η οδηγία. Πρόκειται όμως για τη διασυνοριακή υπερίθαλψη. Αυτό αναφέρεται στον τίτλο και συγχρονίζει ε, ε, την 1408 που είναι ιδιαίτερα απαρχαιωμένη και σε αντίθεση με την νομολογία του 10. Ό,τι και να κάνουμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πω ότι οι ασθενείς έχουν δικαιώματα και θα δικαιωθούν, δεν χρειάζεται να βρεθούν ενώπιον ενός δικαστηρίου. Θα πρέπει να λάβουν επίγουσα περίθαλψη και ακόμα και αν βρίσκονται στο εξωτερικό θα πρέπει να τους αποδίδονται τα έξοδα νοσηλείας όπως και στη χώρα όπου είναι ασφαλισμένη Σε σχέση με τα νοσοκομιακά νοσήλια, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα δαπανηρό εγχείρημα και ο ασθενής θα πρέπει να αποτανθεί στο δικό του κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα να δει κατά πόσο θα του αποδοθούν τα έξοδα. Και στις χώρες ε, προέλευσης δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη κάλυψη. Άρα τα πρόσωπα, οι πολίτες που ταξιδεύουν θα πρέπει να μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην ε, περίθαλψη και όχι μόνο όταν μιλάμε για επίγοντα περιστατικά. Εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία της κυρίας Βερνιό και θα πρέπει να μας δώσει το κράτη-μέλη ορισμένους ποιοτικούς δείκτες για να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα της περίθαλψης. Γιατί εδώ ερχόμαστε σε ρήξη με την επικουρικότητα και γι' αυτό αναρωτηθήκαμε γιατί πρέπει να υπάρχει νομική βάση. Αν πρόκειται για σύσταση θα πρέπει να την συντονίσουμε. Γι' αυτό ζητάμε ποιοτικούς δείκτες για να φτάσουμε σε ένα κοινό συμβιβασμό. Και έτσι εμπλουτίζουμε τον κανονισμό 1408. Δεν θα καταχραστώ άλλο του χρόνου σας. Κυρία Γκέπχαρτ, θέλετε να επανέλθετε, η κυρία Σάλντεμός μετά. Ναι, επιθυμώ να επανέλθω. Γιατί είναι προφανές ότι δεν κατανόησε καλά τα λόγια μου η κυρία Γιώργενσεν. Δεν είπα σε καμία περίπτωση να κάνουμε εκ νέου παραπομπή της οδηγίας στην ε, οδηγίες. Αντίθετα, τη θεωρώ απαραίτητη, διότι σε πολλές χώρες μέλη είναι προβληματική κατάσταση με τα δικαιώματα των ασθενών και όχι μόνο στα όσα προβλέπει τις αποφάσεις του το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα μπορούσα να πω, εντάξει, δεν ανησυχώ τόσο πολύ, διότι στην Γερμανία έχουμε ήδη εφαρμόσει το εθνικό δίκαιο το περιεχόμενο των αποφάσεων του ΔΕΚ. Θα μπορούσα να πω ότι αφού στην πατρίδα μου τα πράγματα είναι εντάξει μπορώ να μην ανησυχώ. Βλέπω όμως και τι επιπτώσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και βλέπω ότι στην Γερμανία τα ταμεία υγεία πληρώνουν θεραπείες πολιτών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Και σωστό είναι αυτό. Σωστό λοιπόν, απολύτω σωστό. Το πρόβλημα που διαπιστώνω ωστόσο ότι υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει με την πάροδο του χρόνου είναι να δούμε επιπτώσεις σε άλλες χώρες μέλη εν προκειμένου. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί Γερμανοί πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν για θεραπείες στην Πολωνία. Για παράδειγμα για, θερα, για θεραπείες ε, οδοντιάτρου. Επειδή λοιπόν οι οδοντιατρικές φροντίδες είναι πολύ φθηνότερες στην, Γερμανία, στην Πολωνία συγγνώμη, από τη Γερμανία είναι προφανές ότι είναι ευνοϊκότερο, φθηνότερο για τους ε, Γερμανούς πολίτες και ασθενείς. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει τώρα όμως στην Πολωνία είναι οι φροντίδες των οδοντιάτρων να αυξάνουν. Ε, συγγνώμη, οι τιμές των οδοντιάτρων είναι να αυξάνουν. Και φοβάμαι πολύ ότι κάποια στιγμή οι Πολωνοί πολίτες που δεν έχουν το ίδιο βιωτικό επίπεδο με τους Γερμανούς δεν θα μπορούν να πληρώσουν πια. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα υπερεπιβαρυνθούν τα πολωνικά ταμεία υγείας γιατί δεν θα μπορούν να πληρώνουν τις υψηλές αυτές τις τιμές. Για μένα αυτό είναι σημαντικό. Και στην περίπτωση αυτή με ανησυχεί το τι θα γίνει με τα δικαιώματα των Πολωνών ασθενών, που και αυτοί πρέπει να έχουν τις ίδιες, την ίδια πρόσβαση στα ίδια δικαιώματα όπως οι Γερμανοί. Δεν θέλω λοιπόν να υπάρξει ένας μη υγιής ανταγωνισμός και γι' αυτό το λόγο πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά. Ποιες επιπτώσεις έχει το, δικαιο, το δίκαιο το οποίο ψηφίζουμε εδώ στα διάφορα συστήματα. Και το άνοιγμα που πάμε να κάνουμε και το οποίο βρίσκω ότι είναι σωστό και το εγκρίνω και θέλω να γίνει πρέπει να γίνει με τρόπο που να λαμβάνουμε υπόψη και το ενδεχόμενο να προκύψουν αντίθετα αποτελέσματα. Τίθετο το θέμα, και το έχει πει και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά επανάληψη, ότι τα συστήματα υγείας των χωρών μελών δεν πρέπει να υπερεπιβαρυνθούν, ούτε πρέπει να αμφισβητηθούν με τα όσα πράττουμε εμεί εδώ. Αυτό ζητώ εγώ. Και όχι μόνο από την σκοπιά των ασθενών εκείνων οι οποίοι είναι ευπορότεροι, αλλά και το τι γίνεται με τα δικαιώματα εκείνων που είναι λιγότερο εύποροι. Και εμείς πρέπει να φροντίσουμε ώστε και αυτοί οι λιγότερο εύποροι ασθενείς να έχουν τα ίδια δικαιώματα στις ίδιες φροντίδες και να μην διευκολύνουμε ένα τουρισμό εντός εισαγωγικών φροντίδων υγείας ο οποίος τελικά θα καταλήξει σε βάρος ορισμένων. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε. Και πρέπει να πούμε ξεκάθαρα να σκεφτούμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι επιπτώσεις, οι συνέπειες της, που νομοθεσίας που ψηφίζουμε εν προκειμένου. Γι' αυτό και λέω ότι πάντα σκεφτούμε τα πράγματα αυτά πολύ προσεκτικά. Και αν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια καλή λύση μέσα στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία, τόσο το καλύτερο. Αν όμως όχι, τότε θεωρώ ότι είναι σωστό να συνεχίσουμε να συζητούμε ίσως για μισό χρόνο παραπάνω. Ίσως τότε εσείς να μην είσαστε εδώ. Κρίμα. Εγώ θα είμαι και στο επόμενο κοινοβούλιο και σας βεβαιώνω ότι ε, θα συνεχίσω να ασχολούμαι με το θέμα. Πάντως θα θέσω υποψηφιότητα και πάλι και ε, θεωρώ ότι θα επανεκλεγώ. Δεν μπορούμε πάντως να εξαρτήσουμε την νομοθεσία από το αν θα είναι ένας συγκεκριμένος βουλευτής εδώ στην επόμενη περίοδο ή όχι, στην επόμενη θητεία ή όχι. Αυτό που απασχολεί εδώ είναι τα δικαιώματα των ασθενών. Όχι μόνο για τούτη τη θητεία αλλά και για την επόμενη. Και αυτό θέλω να πω. Um, Πρόεδρος. Δεν μας οδηγεί πουθενά αυτή η συζήτηση. Κυρία Ντεμόζερ. Να πω στην κυρία Γιώργενσεν το εξής. Νομίζω ότι επίτηδες δεν κατάλαβες, δεν ήθελες να καταλάβεις. Και αυτό μας δίνει κάποια μηνύματα σχετικά με την θέση της ομάδας σου για το ζήτημα των δικαιωμάτων ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι τροπολογίε ε, μεταφρασμένες και να δούμε μετά κατά πόσο θα χρειαστεί να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα ή όχι. Πρόεδρος, να πω και εγώ μερικά πράγματα γιατί έχω καταθέσει καποιε τροπολογιε Σε έχω καταθέσει σε έναν τομέα που θεωρώ ότι ως Επιτροπή έχουμε κάτι να πούμε διότι η πρωτη Κομισιόν είναι κάπως αδύναμη και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα, η ασφάλεια ε, τα πρότυπα ενημέρωση κλπ. Διάβασα σε μια κυριακάτικη εφημερίδα πολλές ε, πληροφορίες και είχε, υπήρχε μια εικόνα της Ευρώπης και οι Άγγλοι ήταν, είχαν αρκετά, ήταν αρκετά προνομιούχοι οι Άγγλοι πολίτες. Και έλεγα επίσης ότι δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ποιότητα, ασφάλεια, προστασία, αν πάτε στο εξωτερικό. Η Κομισιόν λοιπόν έχει συμπεριλάβει στο πλαίσιο της, των προφορίων που χορηγεί αυτά τα στοιχεία και πιστεύω ότι ο πολίτης βρίσκεται σε αδύναμη θέση δεδομένου του ότι στην ε, πρόταση περιλαμβάνουμε κάποια στοιχεία πολύ πιο θετικά από αυτά που έχει θέσει η Κομισιόν ως βάση την πρότασή της. Υπάρχουν πολλά ζητήματα για το οποίο είναι υπεύθυνο. Εγώ διαφωνώ ότι δεν πρέπει να είναι υπεύθυνο το κράτο μέλος το οποίο δεν χορηγεί την θεραπεία, την ενημέρωση που να την παρέχει το κράτο μέλος το οποίο χορηγεί την θεραπεία. Και εδώ νομίζω ότι η Κομισιόν σφάλει. Όχι ότι δεν μπορεί να ρυθμιστεί το ζήτημα, αλλά το πρόβλημα που έχουμε την πρόταση είναι ότι η πρόθεση είναι καλή και πρέπει να συμμορφωθούμε με την απόφαση του 10, αλλά η πρόταση έχει καλές προθέσεις, αλλά μέχρι εκεί. Το ζήτημα δεν είναι κατά πόσο το θέμα θα ρυθμιστεί πριν ή μετά τις εκλογές. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να καθυστερήσει το ζήτημα, άλλοι που θέλουν να επιταχυνθεί. Πάντως το θέμα είναι πολύ σημαντικό, ούτως ή άλλως, και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά, θα πει προς όφελος του πολίτη. Νομίζω ότι είναι δυνατόν να το πετύχουμε, αλλά δεν χρειάζεται να βιαστούμε υπερβολικά. Και όλο τα λέω αυτά είναι πως η Κομισιόν γνωρίζει ότι έχουμε ήδη το ευρωπαϊκό σύστημα υγείας που λειτουργεί. Αν λοιπόν είστε στο εξωτερικό, δικαιούστε νοσηλείας ε, και περίθαλψης. Ούτως ή άλλο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Άλλοι μπορεί να είναι ασφαλισμένοι, άλλοι όχι. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι πολλοί συμπολίτε μου μεταβαίνουν στην Ισπανία, ασθενούν εκεί, φτάνει το ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο του μεταφέρει σε μια κλινική ιδιωτική και πληρώνουν το μέλλον κεφαλά τους. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προβλέψουμε μια καλύτερη ρύθμιση. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε το κείμενο μέσω τροπολογιών. Αλλά πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα νομική ε, ε, ε, ασφάλεια δικαίου, συγγνώμη, και πρέπει να θυμίσουμε και το θέμα της προηγούμενης έγκρισης. Μίλησα με τον δικηγόρο μου που είναι φιλελεύθερος κυρία Γιώργενσεν και είναι υπέρ μιας παρόμοιας πρότασης αλλά επειδή γνωρίζει τις υπηρεσίες υγείας, γνωρίζει και τη χρηματοδότησή τους είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη εξοδότηση από τον αρμόδιο ε, επίτροπο της περιοχής που διαχειρίζεται τα κονδύλια του συστήματος ασφάλειας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός είναι ο οποίος ε, αποφασίζει κατά πόσο θα είναι σε θέση το σύστημα να καταβάλει τα ποσά Το... Η οδηγία αυτή θέλει να πει στον πολίτες ότι μπορείτε να μεταβείτε οπουδήποτε επιθυμείτε για θεραπεία κλπ. Αλλά δεν είναι αυτή η πρόθεση της απόφασης ε, του δικαστηρίου. Βασίστηκε αυτή η απόφαση στην ελεύθερη διακίνηση και πρόσβαση στις υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να μην δώσουμε υπερβολικές προσδοκίες στους ε, συμπολίτες μας ε, πριν από τις εκλογές. Πολλοί ηλικιωμένοι δεν θέλουν να μεταβούν ε, χάρη σε μια λοδαπή χώρα για να τύχουν περίθαλψης. Μ' αρέσει η ιδέα αυτή τη καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα δίκτυα των εμπειρογνωμόνων. Έχουμε εξαιρετικού εμπειρογνώμονε, εξαιρετικά νοσοκομεία και κλινικέ ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω καταθέσει λοιπόν πολλέ τροπολογίε, ειδικά στον τομέα τη ε, ασφάλεια και της προστασίας ε, των πολιτών. Εάν κοιτάξετε λοιπόν την περιπλοκότητα του ζητήματος και του συστήματος, του συστήματος μόνο που υπάρχουν στα κράτη μέλη, η περίθαψη νοσοκομιακή διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Και θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό νομοθέτημα αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κύριε Μπέργκ. Ζητώ συγγνώμη γιατί έπρεπε να ψηφίσουμε στην ΑΦΕΤ. Είμαι σκιώδη σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κινηθούμε προς τα μπρος, να εστιάσουμε την προσοχή μας στον ασθενή σε σχέση με άλλα ζητήματα όπως έχω έχω προναφέρει. Εγώ είμαι δικαιούχος της διασυνοριακής ε, περίθαλψης και εκεί που υπάρχει καλύτερα σε μια χώρα σε σχέση με μια άλλη θα πρέπει να βελτιωθεί. Δεν θα πρέπει να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο τον ασθενή. Μίλησα με ενδιαφερόμενος. Προσπαθώ να περάσω καλές ιδέες αλλά θα πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί γιατί διαφορετικά δεν θα περάσει τίποτα. Υπάρχουν πολύ καλές προτάσεις και θα πρέπει να κινηθούμε σχετικά γρήγορα. κυρία Γιώργενσε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο σημαντικότερο στους ασθενείς. Ως προς τον οδοντίατο στην Πολωνία αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ε, κινητικότητα. Εσείς ε, μιλήσατε για ένα συγκεκριμένο γιατρό και είπατε ότι στην περίπτωση του liberal doctor μπορεί να υπάρξει πολύ υψηλό κόστος. Ένα κράτος μέλος πρέπει να παρέχει περίθαλψη στους κατοίκους του και αν πάει στο εξωτερικό τότε θα του επιστραφούν τα έξοδα, το ισόποσο μάλλον, που θα του στήχιζε στο κράτος μέλος. Άρα πρόκειται για υψηλό ποσό. Άρα υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής. Λέμε ότι υπάρχει πολύ υψηλό κόστος Δηλαδή τι λέμε, να πάνε στην Αλοδαπή 10 ή 20 ας πάνε στην Αλοδαπή. Μα το ποσό μπορεί να είναι το ίδιο, δηλαδή το ισόποσο μπορεί να είναι το ίδιο. Δηλαδή πού να πάει, να πάει στο εξωτερικό για να πεθάνει. Κύρια Γιώργενσεν, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την καλύτερη εμπειρία αποστολή στο εξωτερικό γιατί είχαμε 20, είχαμε 20 χρόνια συντηρητικούς που δεν επένδυσαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα εξάγουμε ασθενείς στη Γαλλία. Αυτό δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι ότι αν ο φιλελεύθερος γιατρός μου είπε είναι φτηνότερο ή ακριβότερο. Απλώς θα πρέπει να βρίσκουμε μια σειρά κριτηρία. Δεν αντιτάχθηκε είπε ότι θα πρέπει να έχουμε ε, λογική προσέγγιση γιατί διαφορετικά δεν ισχύει και ο... δηλαδή μειώνεται και ο εθνικός υπροεπολογισμό. Ίσως είναι λιγότερο δαπανηρό να τους στείλουμε στο εξωτερικό και γι' αυτό και τους αποστέλουμε. Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ιατρική περίθαλψη και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μα γι' αυτό ακριβώς ε, γίνεται αυτό. Γιατί ήταν δυσανάλογο, δυσανάλογο ακριβό να είναι κανείς σε μία λίστα αναμονής. Το ζήτημα είναι ποιος αποφασίζει για το πού θα πάει ο ασθενής. Μιλάμε για προγενέστερη έγκριση. Δεν διαφωνούμε. Το ζήτημα είναι πώς έμπρακτα θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Να μπορεί να μεταβεί ο ασθενής και να μην υποσκάπτουμε το εθνικό σύστημα. Και αυτό αποζητά και η Επιτροπή. Η κυρία Βάιλερ θέλει να επανέλθει. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω λίγα λόγια ακόμα για την αντικειμενικοποίηση, διότι Πρόκειται για κανθόδη κατάσταση σε πολλές χώρες από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ελλάδα. Όλες οι ε, απόψεις που ακούστηκαν είναι σωστές. Πράγματι η ποιότητα των συστημάτων υγείας στις διάφορες χώρες ποικίλει. Είναι γεγονός και είναι και διαφορετικά τα κονδύλια που δαπανούν οι χώρες μέλη για τα συστήματα υγεία τους και για την περαιτέρω εκπαίδευση κατάρτιση του προσωπικού και ιδιαίτερα για ορισμένες δύσκολες νόσους και ασθένειες που μπορεί να είναι η θεραπεία τους εξαιρετικά δαπανηρή. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν μήπως και απαλλάξουμε των ευθυνών τους ορισμένες χώρες μέλη όπως έκανε ίσως η Βρετανία διότι δεν ήθελαν αλλά και που από άποψη ικανοτήτων τους δεν μπορούν. Αμφισβητώ ότι μια χώρα όπως η Λιθουανία για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα τώρα, οι άλλες μικρές χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν τέτοια επιστημονική γνώση για την αντιμετώπιση ορισμένων δύσκολων και περίπλοκων νόσων όπως μπορούν ενδεχομένως κάποιες βιομηχανικές χώρες όπως η Ισπανία, η Γερμανία ή η Σουηδία. Πρέπει να βρεθεί κάποια ισορροπία. Για μένα είναι σημαντικό οι γυναίκες στην Πολωνία άκουσα συγκεκριμένα το παράδειγμα αυτό που αντιμετωπίζουν καρκίνο του μαστού πράγμα το οποίο θεραπεύεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πεθαίνουν οι γυναίκες όμως από το καρκίνο του μαστού στην Πολωνία. Εμείς αναμένουμε από την νομοθεσία αυτή να οδηγεί σε βελτίωση των φροντίδων υγείας. Όχι τώρα να απομονωθούν οι ε, Πολωνοί και να πούν «Α, στο μέλλον όλα αυτά τα πράγματα να τα αναλάβουν οι Σουηδοί και οι Γερμανοί». Αλλά να αναπτύξουν αντίθετα την ικανότητα να θεραπεύουν και αυτή την νόσο η οποία πια έχει γίνει ε, είναι εξαιρετικά εκτεταμένη. Να μην φτάσουμε δηλαδή κάποιες χώρες μέλη να πούν αφού έτσι και αλλιώ έχουμε αυτόν τον τουρισμό φροντίδων υγείας. Μπορούμε τον τάδε ασθενή να τον στείλουμε εκεί και τον άλλο εκεί. Και δεν χρειαζόμαστε καν κέντρα υγείας στα χωριά. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και με τις Εθνικές Βουλές γιατί και αυτές ενδιαφέρονται ώστε και στην τελευταία γωνιά της Λαπωνίας ή σε εμάς στα βαβαρικά δάση να υπάρχει δυνατότητα να προσφερθούν φροντίδες υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερες ανταλλαγές μεταξύ μας ή ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής που υπάρχουν παντού και στη Γερμανία υπάρχουν και να μειώσουμε και τα έξτρα κονδύλια που δίνονται ε, καμιά φορά με τον τρόπο αλλά νομίζω ότι όλες οι χώρες δεν έχουν κάνει επαρκή προσπάθεια για να εξυγχρονίσουν τα συστήματα υγείας των και δεν εννοώ μόνο τη Μεγάλη Βρετανία εδώ, εννοώ και την Γερμανία, δεν το έχει πράξει αυτό. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, έφτασα με καθυστέρηση, αλλά συζητούσαμε το θέμα σε άλλες επιτροπές όπου είμαι σκιώδης θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα. Εμεί είμαστε Επιτροπή ΙΜΚΟ και ακόμα και αν κάποιοι συνάδελφοι τη δεξιά λένε ότι θα πρέπει να έχουμε τι ε, τιμέ ε, που υπάρχουν στην αγορά. Και φέρω εδώ το παράδειγμα τη ε, Ρουμανίας διότι αυτό συμβαίνει συχνά. Υπάρχει πόλωση της κοινωνίας από οικονομικής κοπιάς Μερικοί έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα, μερικοί όχι. Δηλαδή δεν είναι σε θέση να ταξιδέψουν διότι το κράτος θα καταβάλει μόνο τα ποσά τα οποία θα δαπανίσει κανείς εντός της χώρας και το κόστος στο εξωτερικό είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι γνωρίζετε. Φυσικά προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους ασθενείς που μπορούν να ταξιδέψουν μπορούν να πληρώσουν το επιπλέον κόστος που απαιτούν που απαιτεί η περιθεψη στο εξωτερικό, αλλά στη Ρουμανία δεν θα υπάρξει με αυτόν τον τρόπο ένα κίνητρο προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίε υγείας και τα χαμηλά εισοδήματα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εγώ είμαι σκιώδης ηγήτρια στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Εμείς, ε, όπως γνωρίζετε, δημιουργούμε τη ζωή, γεννάμε. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε να έχουμε και κάποια με ευτήρια εγγύς των περιοχών στις οποίες ε, ζούμε. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα να χρειαστεί να μεταβεί στην Αλβαπή για να αποκτήσει το τέκνο της. Υπάρχει και μια πτυχή που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αν κάθε κράτος καταρτήσει έναν κατάλογο με τις ε, υπηρεσίες ε, που παρέχει, θα υπάρξουν προβλήματα στην περίπτωση επιστροφής εξόδων τα οποία έχουν καταβληθεί σε άλλη χώρα. Η οδηγία λοιπόν θα πρέπει να διευκρινίσει όλες αυτές τις παρανοήσεις διότι κάποιο άλλο κράτος να μην συμπεριλαμβάνει την ίδια θεραπεία για την ε, ίδια ασθένεια. Και αυτό αποβαίνει εις βάρος του πολίτη. Πρέπει λοιπόν να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά τα ζητήματα, ειδικά στην δική μας Επιτροπή. Αυτές οι οικονομικές διαφορές ε, που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη χρειάζεται να την υπόψη. Πολλοί γιατροί και πολλοί νοσηλευτές έχουν ήδη εγκαταλείψει την χώρα μου, έχουν μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει έλλειψη ε, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν θέλω να επιμείνω, όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση και έχουμε όλοι υποβάλει τροπολογίε και θεωρώ ότι με την εξέταση των υπολογιών μπορούμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Ευχαριστώ. Θα κλείσω τη συζήτηση στο σημείο αυτό. Είχαμε μια εκτεταμένη συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων κλπ. Δώσω το λόγο στην εισηγήτη. Δεν ξέρω η Κομισιόν θέλει να προσθέσει κάτι. Σας είδα να ε, ε κάνετε πολλέ γκριμάτσες όταν ε, μίλαγα ειδικά εγώ να μου πείτε τι πρόβλημα υπήρξε. Δεν θα μπορούσα να πω φυσικά ότι σφάλετε, αλλά θα θέλω να ευκνήσω κάποιες πτυχές. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η πρότασή μας ε, προετοιμάστε και μετά από πολύχρονο, ε, πολύχρονο προβληματισμό και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα ορθολογική ε, διευκρίνηση των δικαιωμάτων των πολιτών τηρώντας το αποφάσεις του ΔΕΚ και προσθέτοντας κάποιες διασφαλίσεις ζητήματα ασφάλειας και προστασίας. Ε, εδώ νομίζω ότι δεν ε, προτείνουμε μια απλή ενημέρωση του ασθενούς. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να λάβουν τη συλλογική πολιτική ευθύνη στο να καθορίσουν πρότυπα ασφάλειας και προστασίας και να διασφαλίσουν τον έλεγχο. Αυτό το ζητάμε λοιπόν, να αναλάβουν λοιπόν αυτή την πολιτική ε, απόφαση δεδομένου του ότι πρόκειται για έναν τομέα ε, πολύ σημαντικό. Θέλαμε λοιπόν να προσθέσουμε αυτήν την ε, εξασφάλιση της ε, παροχής περίθαψης στους ασθένει Μερικές παρατηρήσεις, η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η οδηγία θέλει να συμπληρώσει τον κανονισμό για την κοινωνική ασφάλιση. Ε, να το συμπληρώσει. Υπάρχει ήδη, ξέρουμε πως υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για την ε, οδηγία αυτή. Η δική μας πρόταση ε, συμπληρώνει, επαναλαμβάνω. Και αυτό δεν σημαίνει επικάλυψη, δηλαδή να επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα προσπαθούμε να τηρήσουμε την νομοθεσία του ΔΕΚ. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος από τον κανονισμό. Εσείς θα πρέπει να τον προσδιορίσετε αυτόν το δρόμο. Τώρα για τις ανισότητες ακούσαμε πολλά να λέγονται από πλευρά Κοινοβουλίου και εμείς η Επιτροπή προσπαθήσαμε να τηρήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των ασθενού και τα συστήματα που ισχύουν στα κράτη-μέλη όπου θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες διότι οι πολίτες δεν έχουν τη διάθεση να μετακινούνται ανά την Ευρώπη για να θεραπευθούν Προσπαθήσαμε λοιπόν να σεβαστούμε αυτές τις ε, αρχές των συστημάτων υγείας, δεδομένων και των δυσκολιών που υπάρχουν στο επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο και ε, προσπαθούμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα των ε, επιστροφών, των και κλπ. Εντάξει, υπάρχουν ισότητε στην Ευρώπη και στο ιστορικό κάθε κράτο μέλους Όλοι δεν έχουν τα ίδια μέσα για ταξίδι, μετακινήσεις κλπ. Ε, το γεγονό είναι ότι εμεί δεν μπορούσαμε σε αυτή την οδηγία να διορθώσουμε τα πάντα, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε και από τα υγεία, να ευνοήσουν την μετακίνηση των ασθενών. Ακούσαμε τις, ε, το ζήτημα των ε, θεραπείας των δοντιών για τις διάφορες πλαστικές ε, εγχειρήσεις κλπ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου για τις ανισότητες, αλλά σας εξηγήσω ότι εμείς θελήσαμε να λάβουμε υπόψη τις, ε, τους δεσμεύσεις και τους περιορισμούς των προϋπολογισμών στα θέματα υγείας. Ακούσαμε επίσης το ζήτημα του ορισμού των ε, νοσοκομιακών υπηρεσιών. Αν έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς ε, καταλόγους, ε, πιο, πώς θα καταλαβαίνει ο ασθενής ε, ποιος είναι ο σωστός κατάλογος, στους πίνακες και θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Κυρία, κυρία Ρόιτοβα, ακούσαμε τις προτάσεις σας, ακούσαμε και άλλες προτάσεις. Πάντως πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο επιθυμεί να αποσαφηνίσει την νομοθεσία ένα κείμενο το οποίο θα είναι απλό και κατανοητό από τον πολίτη, να μην έχουμε 27 συστήματα τα οποία θα δημιουργούν δυσκολίες στην κατανόηση από τους πολίτες. Η κυρία Βερνιό, θα λάβω το λόγο. Εγώ μη με παρεξηγείτε, δεν είπα ότι έχουμε μόνο μία οδηγία κοινωνικής ασφάλισης. Εγώ είπα ότι καταρχήν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για επίγουσες περιπτώσεις πρέπει να είναι σαφές, αλλά δεν είναι λειτουργικό. Επί χάρτου είναι πολύ καλό, αλλά έμπρακτα είναι δύσκολο. Και πάντα βρίσκουμε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο σε αυτήν την Επιτροπή, η μεταφορά και εφαρμογή. Κύριε Βερνιό. Ευχαριστώ. Πώς να ανακεφαλαιώσω ένα θέμα που δημιουργηθεί τέτοια πάθη. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε σε... Αντιμετωπίζουμε ένα πολύπλοκο ζήτημα. Είχαμε πληθώρα συζητήσεων. Διαπιστώνω και αυτό με ευχαριστεί γιατί υπάρχουν πολλά εκρεμή ζητήματα τα οποία είναι άκρος ανησυχητικά. Με ευχαριστεί όμως ότι η, ομάδα της, η σοσιαλιστική ομάδα έχει μία σαφή κατευθυντήρια γραμμή και αυτό με καθησυχάζει διότι ποτέ δεν ετέθη ζήτημα αντίθεση σε αυτή την οδηγία. Εμείς ψηφίσαμε να υπάρξει μια οδηγία που να ε, διασαπίζει τα δικαιώματα των ασθενών. Άρα όλοι λέμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών χωρίς να απο Κλείσουμε μια κινητικότητα όταν είναι αναγκαία. Η Μπάρμπαρα τόνισε ορισμένες περιπτώσεις και παράλληλα χωρίς να θέλουμε να φτάσουμε σε έναν ιατρικό τουρισμό που θα οδηγούσε στα προβλήματα που τόνισε η Εύλην μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας. Ε, και εμείς έχουμε πρόβλημα στον ε, οδοντιατρικό τομέα και δεν μιλάμε για αισθητικές επεμβάσεις το έχουμε εμεί το πρόβλημα με την Ουγγαρία. Δηλαδή, ορισμένες χώρες απομακρύνονται από τις ευθύνε τους. Ε, λυπάμαι που ο κύριος Σφάμπ δεν είναι εδώ. Μίλησε για καταναλωτές. Αυτό με σοκάρει, γιατί δεν καταναλώνουμε... Ε, δεν μιλάμε για καταναλωτισμό ή κατανάλωση όταν μιλάμε για ιατρική φροντίδα. Εδώ πρόκειται για ασθενείς και το κείμενο της Επιτροπής. Αν και περιορισμένο, δεν είναι ικανοποιητικό. Και αυτό το αποδεικνύει η συζήτηση. Πολλά πράγματα πρέπει να αποσαφινιστούν. Θα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοοικονομική εξισορρόπηση, όπως είπε η Ζωέλ, ανάλογη με την περίθαλψη. Γιατί αν υπάρξει ε, έκρηξη και καταράκωση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης αυτό θα είναι ολέθριο. Μιλάμε για κινητικότητα των ασθενών. Ας λάβουμε υπόψη βεβαίως και τους επαγγελματίες, η Γκαμπριέλα το τόνισε, γιατί οι πολιτικοί θα πρέπει να έχουν ένα όραμα, ένα πολιτικό που υπερβαίνει τη μία γενιά, όπως έκανε ο Ζακ Ντελόρ. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ως προς την ρύθμιση των μείζων ζήτημάτων που υπάρχουν σε αυτό το κείμενο που δεν αποσαφηνίζονται από την Επιτροπή. Χρειάζεται χρόνος, όλοι συμφωνούμε. Λυπάμαι που έφυγε ο κύριος Σβάμπ γιατί είπε ότι ζητήσαμε αργά την έκθεση εμπειρογνωμόνων και η κυρία Μακάρθη και η συντονίστρια από το Φθινόπωρο ζήτησε αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των τριών επιτροπών της ε, ΕΜΒΗ, ε, της, του περιβάλλοντος και της ΙΜΚΟ. Και χαίρομαι διότι επιμείναμε. Έτσι στις 3 Μαρτίου θα έχουμε μία έκθεση νομικού περιεχομένου. Θα γίνει μια συνάντηση με όλους τους σκιώδεις την επόμενη πέμπτη γιατί υπάρχουν κοινά σημεία. Συμφωνώ με ορισμένα σημεία που έφυξε η κυρία Ρόιτοβα. Υπάρχει ένα κοινό πεδίο, μιλάμε για ποιότητα, ασφάλεια, δικαιώματα ασθενών χωρίς να καταδικάζουμε τα εθνικά συστήματα υγείας και να τα θέτουμε σε κίνδυνο. Θα πρέπει να περιμένουμε τώρα τη γνωμοδότηση της νομικής επιτροπής να μας προτείνουν μια νομική βάση. Άρα Στρασβούργο για να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Και ελπίζω ότι έτσι σας δίνουμε και λίγο περισσότερο χρόνο για να συζητήσετε με τους καταθέσαντες τις τροπολογίες. Δεν θα είναι εύκολη η διαδικασία. γιατί έχουμε περίπου 1.400 τροπολογίες σε διάφορες επιτροπές, 700 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και το καθεξής. Θα είναι λοιπόν ε, πολύ δύσκολη η διαδικασία μέχρι ότου η συνένεση του Κοινοβούλιο. Πρέπει να γίνουν και άλλες συζητήσεις και ελπίζω εσείς κύριε να μην αισθανθήκατε ότι σας παραφορτώσαμε εμείς οι γυναίκες σήμερα. Α, είσαστε πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ωραία. Δεν αντιμετωπίζω καμία δυσκολία. Θεωρώ όμως, κυρία Πρόεδρε, να μην, ε, είναι σημαντικό να μην χάσουμε το στόχο από τα μάτια μας. Να μην μπούμε δηλαδή σε μια πολιτική διαμάχη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. έχω εντονότατο ενδιαφέρον για να λάβουμε τις σωστές ε, αποφάσεις. Εγώ δεν ασχολούμαι, δεν ε, ε, προωθώ καμία πολιτική, οι πολιτικές ομάδες θα κάνουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει όντως να κάνουμε σωστές διαδικασίες. Είναι σωστό να λειτουργήσει εν τέλει η οδηγία. Νομίζω ότι όντως χρειαζόμαστε οδηγία στον τομέα αυτό και να υπάρξει νομική ασφάλεια και σαφήνεια Στα 15 χρόνια που είμαι ευρωβουλευτής είδα καμιά φορά να απαιτείται βελτίωση των ε, προτάσεων της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ όλες και όλους.